συμφωνία που διαπραγματεύεται μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή τακτική έξοδος, και τρίτον, τι θα γίνει σε περίπτωση άτακτης εξόδου. Πάμε λοιπόν συγκεκριμένα στο σημείο 4. Είχαμε για έκτη φορά μία δημοσίευση ε, ετοιμότητος της ε, Κομισιόν για την, για την περίπτωση του Brexit. Και, λέει υπό το φως της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας γελάω γιατί είναι το, το ελάχιστο μπορεί να πει κανεί. Τέλο πάντων, τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την ε, τακτική έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, τέσσερις Σεπτεμβρίου υπέβαλε ένα τροποποιημένο ψήφισμα σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να αναλυθούν τον τομέα της αλληλείας. Μέχρι και το έτος 2020 των μέτρων ετοιμότητας που ήδη εφαρμόζονται για την ε, πρόσβαση των ευρωπαϊκών σκαφών στα βρετανικά ύδατα και των βρετανικών στα ευρωπαϊκά οι συντονιστές προηγουμένως συζήτησαν μια απλουσταμένη διαδικασία χωρίς τροπολογίες σύμφωνα με τον κανόνα 22, 52 ε, με συγχωρείτε, και εγώ ως πρόεδρος θα υπέβαλα την τροποποιημένη νομοθετική απόφαση την ερχόμενη εβδομάδα μετά την συζήτηση που σίγουρα θα έχουμε. σε αυτό το σημείο νομίζω ότι μπορώ να δώσω το λόγο στην Κομισιόν για να μας εξηγήσει την πρόταση. Ο κύριος Γιούστα Κούπα. Παρακαλώ. Και ο συνάδελφός σας, κύριος Μπίλιετ, α, δεν είναι εδώ. Ο κύριος Κούπα. ευχαριστώ. Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Με μεγάλη χαρά συμμετέχουμε στην συζήτηση αυτή πρώτο και τρίτο σημείο από αυτά που αναφέρετε είναι ε, ομοιάζουν αρκετά, δηλαδή για άτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα μείνω όμως το πρώτο, υπό την έννοια ότι έχουμε μία πρόταση επιτάπητος και αν μου επιτρέψετε θα γυρίσω λίγο πίσω στον χρόνο και κάποια που του συναδέλφου από τα μέλη του Κοινοβουλίου δεν ήταν εδώ όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση αυτή και θα δώσω ε, ε, λίγο πλαίσιο. Εδώ. Ο κανονισμός ε, για την βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων είχε υιοθετηθεί προκειμένου να διαφολύνει κάθε είδους αλληλευτική δραστηριότητα στα ύδατα άλλων κρατών Εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς συμφωνίες. Υπάρχουν πέντε διαφορετικές δηλαδή αν θέλετε πλαίσια διαδικασίας ή ε, εντός των οποίων μπορεί να γίνει αυτή η χωρι συμφωνιε υπαρχουν πεντε διαφορετικες δηλαδη αν θελετε πλαισια διαδικασια η εντος των οποιων μπορει να γινει αυτη η δραστηριοτητα Και τότε βεβαίω δεν είχαν ληφθεί υπόψη, ε, ε, υποψίες ή περιπτώσεις τύπου Brexit, κανείς δεν το υποψιαζόταν τότε. Τώρα λοιπόν υποβάλλουμε μια τροπολογία τροποποίηση του κανονισμού αυτού ή στο πλαίσιο της προετοιμασία, ε, προετοιμασίας, της δηλαδή έναντι τέτοιων ενδεχομένου. Περιμένουμε να έχουμε μια συμφωνία και επομένως ε, μη άτακτη αποχώρηση αλλά καθώς ε, πλησιάζαμε την προηγούμενη προθεσμία 29 Μαρτίου είχαμε προετοιμάσει ένα σχέδιο τιμότητος με άτακτη αποχώρηση. Και προτείναμε λοιπόν δύο συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Καταρχά το πι θα επανέλθω. Και για τον τομέα τη για την βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών λοιπόν στόλων, που είναι ΣΜΕΦ ως ακρόνιμο. Στο ΣΜΕΦ λοιπόν δεν υπήρχε κάποια διευκόλυνση, κάποια δυνατότητα πρόσβασης για τα βρετανικά σκάφη στα ευρωπαϊκά ύδατα και αντίστροφα για τα δικά μας σκάφη. Αυτό έλειπε και θέλαμε να εισαγάγουμε αυτήν τη δυνατότητα. Και θα πω με σαφήνεια, αυτή η τροποποίηση δεν εισάγει αμοιβαία πρόσβαση, αμοιβαία δυνατότητα πρόσβασης. Είναι μία λύση για την δυνητική περίπτωση να έχουμε άτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε τεχνικώ να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης, δηλαδή να έχουν τα σκάφη όλα τα έγγραφα που θα του χρειάζονται, τις άδειε πρόσβασης. Αλλά να μην γίνει καμία παρανόηση. Δεν μιλούμε για αμ, αμοιβαία δραστηριότητα ή πρόσβαση. Αυτό το χειρίζεται η Συμφωνία Αποχώρησης και θα το χειριστούμε στις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για τεχνική διευκόλυνση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα σκάφη θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ύδατα έχοντας μαζί τους τα κατάλληλα έγγραφα, πιστοποιητικά. Το χρονοπλαίσιο όμως ήταν αρχικά ένα έτος μόνο από την πρώτη προθεσμία. Τώρα που είχαμε την προέκταση μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αντιμετωπίζουμε μια δυνητική περίπτωση να μην έχουμε αποχώρηση 1η Νοεμβρίου και θα πρέπει να δούμε και πέραν αυτού εντός του 2020 και προτείνουμε ένα σχέδιο τιμότητας για το 2020. Τι προτείνουμε. Τρία τινά Αφενός ο κανσμός ΣΜΕΦ της διαχείρισης των εξωτερικών στόλων να επιτρέπει fast track διαδικασίες αδιαδότησης για τα ευρωπαϊκά σκάφη για την ελήψη σε βρετανικά ύδατα. Fast track λοιπόν για τα ευρωπαϊκά σκάφη να μην χρειάζονται να περιμένουν μία, δύο, τρεις, τέσσερις εβδομάδες. Η πρόσβαση στα βρετανικά ύδατα θέλουμε να είναι όσο πιο ταχεία θα γίνεται και συμπεριλαμβάνουμε επέκταση στο ΣΜΕΦ τη τροποποίηση για την αντίστοιχη πρόσβαση των Βρετανικών σκαφών στα δικά μα ύδατα. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Και ένα τρίτο στοιχείο που ε, επεκτείνεται είναι η ανταλλαγή ποσοστώσεων. Δεν έχουμε τέτοιο είδους παράδοση το έχουμε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχουμε με τρίτα κράτη. Έχουμε μια διευκόλυνση ανταλλαγή ποσοστώσεων με το Ηνωμένο Βασιλείο, κατά τρόπον ώστε να είναι όλοι καλυμμένοι εντό του χρονικού πλαισίου προβλέπεται. Πρόκειται για μια τροποποίηση επέκταση της προηγούμενης τροποποίηση που είχε εγκριθεί το 2019 και για όλο το έτος 2020 για να διευκολυνθεί με η αδειοδότηση και, και επαναλαμβάνω δεν μιλούμε για αμοιβιότητα. Και υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο ότι σε όλο αυτό το θέμα των αδειοδοτήσεων πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα κριτήρια βιωσιμότητας του κανονισμού ΣΜΕΦ και ότι αυτά θα τηρούνται. Και υπάρχει μια διαφορά από πέρυσι όταν είχαμε συμφωνία στα τάκ και ποσοστώσεις ως θεμέλιο αυτής της βιωσιμότητας με το Ηνωμένο Βασιλείο να είναι παρόν στη διαδικασία λύσης απόφασης αλλά δεν έχουμε εγγυήσει ότι το 2020 αν έχουμε άτακτη αποχώρηση θα έχουμε συμφωνία τάκ και ποσοστώσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι εκδίδοντα τι άδειε. τις θα εκπληρούνται οι δοκιμές βιωσιμότητας. Και η τροποποίηση αναφέρεται και σε αυτό. Κατά τα άλλα είναι ακριβώς το ίδιο που είχαμε κάνει και την Άνοιξη. Νομίζω ότι προς το παρόν αυτά θα μπορούσα να σας πω. Ευχαριστώ για διευκρίνηση. Δεν διάβασα πουθενά στην έκθεση αν υπάρχει ένδειξη για το τι λέει Βρετανική κυβέρνηση ή αν λέει κάτι Βρετανική κυβέρνηση. Δηλαδή, ουσιαστικά από τη μία πλευρά μόνο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνεται η έγκριση αυτής της παράτασης για τα αλλιευτικά σκάφη να μπορούν από το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή να αλλιεύουν στην Ένωση αν υπάρξει ε, η αμοιβότητα. Αλλά η απάντηση της ε, Βρετανικής κυβέρνησης ποια είναι και κάτι ακόμη για το UN Clause, ε, για το δίκαιο της θάλασσας, τη Διεθνή Σύμβαση. Υποχρέωση συνεργασία στη διαχείριση κοινών αποθεμάτων. Υπάρχει αυτή η διάταξη. Και το δεύτερο, η ανάγκη ελαχιστοποίησης οικονομικών, ε, οικονομικής διαταραχής ή αναταραχής. Γιατί εδώ μιλάμε πλέον για μια νέα αποκλειστική οικονομική ζώνη. Στην πράξη αυτό πού μας οδηγεί. Δηλαδή, τα ενωσιακά σκάφη που ιστορικά αλλιεύουν στα ύδατα δυνάμει της σύμβασης μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν ή όχι. Δεν φαίνεται να ισχύει πια αυτό. Ε, τι έχετε να μας πείτε απάντηση για το πρώτο σημείο. Ποια είναι η απάντηση του Ηνωμένου Βασίλειου. Ρωτήστε το Ηνωμένο Βασίλειο, τέλο πάντων. Εμεί, ίσω να μην το είπα ξεκάθαρα, εμεί θέλουμε από δική μα πλευρά όλα να είναι έτοιμα για να υπάρχει αμοιβαία πρόσβαση στα ύδατα που να λειτουργεί. Και υποθέτουμε ότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο πράγματι συμφωνεί δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει αυτή η αμοιβαιότητα. Άρα αντίστοιχε προετοιμασίε πρέπει να κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά δεν θέλω να κάνω εικασίε. Είπε ότι θα απαντήσει. Ε, μάλλον είπε ότι θα ακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρο της νομοθεσίας. Αλλά δεν μπορώ να αρχίσω να φαντάζομαι τώρα τι μπορεί να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμεί θέλουμε να προετοιμαστούμε για αυτό το ενδεχόμενο να έχουμε πρόσβαση στα δικά του ύδατα, αν μα τα διαθέτουν. Αλλιώ, αν δεν είμαστε έτοιμοι, δεν μπορούμε να στείλουμε σκάφη. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχα και διευκόλυνση για τη δική του την πλευρά, αν δηλαδή εμεί ανοίξουμε τα χωρικά μα ύδατα για αυτού, πάλι δεν θα είναι εύκολο. Δηλαδή, εμείς ετοιμαζόμαστε από τη δική μας πλευρά για το ενδεχόμενο ενός άτακτου Brexit και αν υπάρχει πρόσβαση στα δικά τους ύδατα. Αλλά feedback δεν έχουμε για αυτή την πρόταση, για την προηγούμενη πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλα αυτά... Α, πρέπει να τα λέω πιο αργά. Ναι. Το 2018 ξεκίνησαν όλοι. Όταν ήμασταν εν μέσω των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση και ο τότε υπουργό τη κυβέρνηση, ή ο υπουργό τη τότε κυβέρνηση, αν θέλετε, είχε πει ότι το 19 θα μπορούσε να μην αφήσει ανοιχτά τα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έχουμε όμως επιβεβαίωση τέτοια για το 2019, μάλλον για το 2020 αν δεν υπάρξει συμφωνία, αλλά τεχνικά εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ένα αυτό. Το δεύτερο, για το Γιούγκλος την υποχρέωση συνεργασία, για την ε, ε, διαχείριση των κοινών αποθεμάτων και για την αλεξιτοποίηση ε, διαταραχών. Πράγματι, τα λέει αυτά η σύμβαση και ελπίζουμε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις διατάξεις. Αλλά το θέμα είναι τι μελλοντικέ σχέσει θα έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, είναι ότι γνωρίζουμε και νομίζω γνωρίζει πολύ καλά το Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιε είναι οι υποχρεώσει, και ελπίζω ότι θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ε, όπως αυτές απορρέουν από το και όταν αποχωρήσουν. Αλλά να μην αρχίσω εικασίες και πάλι. Αλλά και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Μάλλον είναι πολύ καλά τα αγγλικά σας. Παρόλα αυτά, είναι τόσο καλά τα αγγλικά σας που δεν ήταν ξεκάθαρα αυτά που είπατε. Εδώ μιλάμε για παράταση ενός καθεστώτος που ισχύει. Και λέτε να ρωτήσω με τη Βρετανική κυβέρνηση. Και λέτε δεν είχατε εσείς feedback. Έτσι δεν λέτε. Δεν είχατε. Και για το Young Μιλήσατε για κάποιες υποχρεώσεις. Engagement και resort obligations. Τι είναι αυτό μπορούμε ή δεν μπορούμε να ψαρέψουμε. Ευχαριστώ για το κοπλιμέντο, για τα αγγλικά που μιλάω. Δεν είπα εγώ στην ίδια πρόταση ότι θα πρέπει να ε, στήσουμε να μας πει το Ηνωμένο Βασίλειο και ότι δεν έχουμε feedback. Είπα, ρωτήστε αν θέλετε να μάθετε την άποψη, αλλά ναι, feedback δεν είχαμε. Ούτε και αντιρρήσεις εφράστησαν όμως από τη δική τους πλευρά στο Συμβούλιο. Στην απόφαση και διαπραγμάτευση έγινε νωρίτερα, ήταν παρόν το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρότι υπήρχε μια χωριστή ομάδα εργασία, οι διαπραγματεύσει έγιναν και στο Κορεπέρ, παρουσία του Ηνωμένου Βασίλειου και εκεί δεν ακούσαμε κάποια ένσταση από βρετανική πλευρά. Αλλά δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για το ότι προετοιμάζονται και δεν μπορώ να κάνω εικασίες περαιτέρω, όπως σας είπα. Για το Γιούγκλος. Δεν είμαι νομικός, μπορώ να λέω καλά, να μιλάω καλά αγγλικά, αλλά δεν είμαι και νομομαθής. Αν δούμε το Γιούγκλος και τα δικαιώματα στα 200 μίλια είναι σαφή. Ένα από αυτά είναι πως ένα κράτος μπορεί να χειρίζεται και τα εχθεαποθέματα, εδώ θα εστιάσουμε, εντός των 200 μιλίων. Όταν ένα απόθεμα είναι κοινό, σε διεθνή είδατε με ένα άλλο κράτος, τότε υπάρχει υποχρέωση αναζήτησης της κοινή συνδιαχείρισης. Η αποχρέωση δεν είναι να καταλήξει αποτέλεσμα, να αναζητήσεις, να προσπαθήσεις να το πετύχεις. Δηλαδή, ναι με να αναζητούμε την κοινή διαχείριση, αλλά δεν είναι υποχρέωση να την πετύχουμε. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, σίγουρα μετά υπάρχει ε, ρύθμιση των διαφορών, αν μία από τις δύο πλευρές δεν τηρεί τις κτλ. Αλλά αρχικά δεν υπάρχει υποχρέωση να βρεθεί μία ε, συμφωνία για τη συνδιαχείριση, αν οι πλευρές δεν είναι πρόθυμες να καταλήξουν συμφωνία. Και αν πράγματι είναι έτσι, θα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και τα κριτήρια της Ούγκλος είναι ξεκάθαρα. Για το τι εφαρμόζεται όταν γίνουν διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και για οικονομικές ε, μετακινήσεις, ε, μεταγκαταστάσεις κτλ. Ε, κτλ. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Αλλά τι είναι engagement, Εδώ είπαμε ότι δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση για να καταλήξουμε σε συμφωνία. On the speaking list, I've got, um, Mr. Van Dalen, uh, Ms. Aguilera, Mrs. Ο κύριος Φαντάλεν, η κυρία Αγγιλέρα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα δεν το γνωρίζει κανείς. με το Brexit. Μπορούμε βεβαίως να το ρίξουμε στον κλήρο, αλλά μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, σε λίγες εβδομάδες, το Brexit θα λάβει χώρα. Και μάλλον χωρίς συμφωνία. Εγώ λυπούμαι, λυπούμαι βαθιά για αυτή την προοπτική, διότι το Brexit μόνο ε, απώλειες θα προκαλέσει και από τις δύο πλευρές της ε, μάχης και από τις δύο όχθες της μάχης. Όπως γνωρίζετε, η πολιτική αλίας είναι ουσιώδου σημασία και για μας και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών διαπραγματεύσεων, συζητήσεων, αφορά όλες τις περιοχές ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Σκοτία, την Ουαλία. Είναι ένα θέμα με ιδιαίτερο οικονομικό βάρος. Υπάρχουν πολλές εταιρείε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία και στις κάτω χώρες που τις πλήττει. Κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους, αλλά Πάρα πολλές εταιρείες θεωρώ ότι ανησυχούν. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να κατεβάσουν ρολά. Ε, νομίζω λοιπόν η κατάσταση είναι, ιδιαίτερη δυσάρεστη, είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πραγματικότητα και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Για αυτά που είπε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να έχουμε απόψη μας την προοπτική ενός σκληρού Brexit χωρίς συμφωνία. Για τα θέματα αμοιβαιότητα στη θάλασσα, λοιπόν, και επειδή τα αναφέρατε, χρειάζεται τεχνική προετοιμασία. Είναι σαφέ ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι από άποψη ε, τεχνική και τεχνοκρατική. Όμω, από την ε, πλευρά τη αμοιβαιότητα, τι θα κάνουμε όταν λέμε αμοιβαιότητα. Σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι οι ψαράδες μας, οι αλείς μας, πρέπει να γνωρίζουν αν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ύδατα ή όχι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη Βόρεια Θάλασσα για τι αλληλευτικέ του δραστηριότητε. Ωραία είναι η τεχνική προετοιμασία, αλλά πώς θα βεβαιωθούμε ότι η αμοιβαιότητα εφαρμόζεται και γίνεται σεβαστή. Πρέπει να εφαρμόζεται και πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και τη δική μας την αλεία και να είμαστε βέβαιοι ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας γίνεται σεβαστή. Πώς θα το χειριστούμε. Πέραν της τεχνικής, πέραν της τεχνικής προετοιμασίας και έχω ξαναπεί, σας ευχαριστώ πολύ για όλη αυτή τη δουλειά, το ζητούμενο είναι να ξέρουν οι αλλοί μας πώς αυτή η αμεβαιότητα θα ισχύσει, πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτή είναι η ερώτηση λότο για μας. Μην ξεχνάμε τι θα μπορούσε να συμβεί αν δεν υπήρχε η αμοιβαιότητα. Θα είναι κάτι πολύ δυσάρεστο. Brexit λοιπόν, με ή χωρί συμφωνία και σε σχέση με αυτό το θέμα. Τι θα μπορούσε να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, κυρία Αγγιλέρα. Mm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεδομένης της περιπλοκότητας και όπως λέει και ο Βαντάλεν ότι δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει αυτό, σε τι θα καταλήξει. Αν έχουμε μία συμφωνία καλώς, αν δεν έχουμε, όλα είναι ανοιχτά. Και αναφέρομαι, μια και είναι εδώ εκπρόσωπος Κομισιόν, σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Αναφέρθηκε εκείνος στη διευκόλυνση της ανταλλαγής ποσοστώσεων αυτό που τώρα έχουμε εντός των κρατών μελών, μεταξύ των κρατών μελών. Και μεταβατικά μέχρι ότου υπάρξει τελική συμφωνία. Αυτή η διευκόλυνση αντιλαμβάνομαι τη στόχευση που θα είναι πάνω απ' όλα να έχουμε μια ομαλή μετάβαση προ της ολόκληρης συμφωνίας, αλλά αυτό μου γύρει κάποια ερωτηματικά. Εάν έχει υπάρξει έξοδος, αυτό θα ισχύσει μέχρι ότου να έχουμε μια αλλιευτική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα. Η επέκταση λοιπόν που αναφέρεται μέχρι το 2020 θα ήταν σε περίπτωση αποχώρησης και αναμένοντας τη νέα συμφωνία, αν κατάλαβα καλά. Γιατί το της ανταλλαγής ποσοστώσεων μου δημιουργεί κάποιες απορίες και ήθελα να καταλάβω αν είναι μόνο αυτό. Τώρα, αντιλαμβάνομαι επίσης την πολιτική βούληση, αλλά είναι δύσκολο τα κριτήρια του κανσμού βιώσιμης διαχείρισης να τηρούνται από αμφότερες πλευρές. Δηλαδή, πώς θα εγγυηθούμε ότι αυτό θα γίνει. Πώς θα είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει δηλαδή τήρηση των κανόνων βιώσιμης διαχείρισης Δεν ξέρω κατά πόσον και η Βρετανική πλευρά θα χρειαστεί μια τροποποίηση νομοθετική δική της προκειμένου να τηρεί τους κανόνες αυτούς. Αντιλαμβάνουμε, ξαναλέω, την πολιτική βούληση να έχουμε αμοιβέ αν θέλετε, διευκολύνσεις να υπάρξει μια ηρεμία και μια ομαλότητα προς τη μετάβαση της σχέσης μας με το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα. Το οποίο μπορεί να διαρκέσει ένα έτος, ένα ενάμεση έτος, λέει ο ομιλήτρια. Αλλά πώς θα εξασφαλίσουμε την τήρηση των διατάξεων των κανόνων αυτών. Πάντως, ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τις τροποποίησεις που υποβάλλει η Κομισιόν και είναι ένα μέτρο εντός του χαοτικού πλαισίου το οποίο δυνητικά αντιμετωπίζουμε να υπάρξει μια ηρεμία, μια ομαλότητα. Mrs. Memory. Κυρία Memory. Όμως συγχωρείτε λειτουργεί. Βλέπω γύρω μου πολλούς ανήσυχους ανθρώπους σε αυτή την αίθουσα. Ο κανονισμός αυτός έχει να κάνει με την αμοιβαία πρόσβαση. Λέτε ότι είναι δίκαιο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Είναι το μέσο που έχετε χρησιμοποιήσει για να κλέβετε τα ψάρια μας. Σας ανησυχεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ότι με τα, στα είδατα αυτά δεν θα έχετε πια πρόσβαση αν δεν υπάρξει συμφωνία για τον Brexit. Ξέρετε όμω τι κοινωνικέ και οικονομικέ απώλειε που έχετε προκαλέσει. Τα αποθέματα ε, ξαντλούνται Ξέρετε, λέτε πως ε, οι στόλοι δεν θα μπορούν πια να ψαρέψουν. Τα ίδια όμως γίνονται και στις χώρες σας. Ε, δείτε τι έχετε προκαλέσει απέναντι. Από την αλληλευτική σας ευημερία πολλά βασίζονται ε, σε αυτά που έχουν πληρώσει ως τίμημα οι βρετανικές παράκτιες κοινότητες. Και πέραν αυτού είσαστε χαρούμενοι και θα θέλετε να παραμείνουν τα πράγματα έτσι. Δεν θέλετε αλλαγή. Δεν θέλετε να υπάρξει συμφωνία, μάλλον θέλετε να υπάρξει συμφωνία αποχώρησης και όχι σκληρό Brexit. Και τα βρετανικά ψάρια θέλουν, ε, οι βρετανικοί αλείς θέλουν ε, συμφωνία. η βρετανία αλείς δεν θα παραχωρήσουν 80% ε, των αλληλευτικών ευκαιριών σε ευρωπαϊκά σκάφη όπως ε, η νομοθεσία για τι εκφορτώσει είναι νομοθεσίε που σε εμά δεν προσφέρουν τίποτα. Έχετε καταλυστεύσει τις φυσικού μα πόρου. και θέλουμε να επιστρέψουν οι προοπτικέ ευημερίε στις δικέ μα παράκτιε κοινότητε. Θέλουμε να στηρίξουμε τη δική μα αλληλευτική βιομηχανία, ψώνοντα τη φωνή τη και κάνοντα την να ακουστεί, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τη σεβαστεί. Ευχαριστούμε, ο κύριο Χάουερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να συμφωνήσω με την κυρία Αγγιλέρα. Όταν είπε ότι θα πρέπει να είμαστε λογικοί στην ε, προσέγγιση μα. Ευχαριστώ την Επιτροπή που όντω υπήρξε λογική και να θυμίσω ότι κάποιοι από εμά στο Ευρωκοινοβούλιο, Βρετανοί βουλευτές, προσεγγίζουμε το θέμα με ψυχραιμία και ορθολογισμό. Μήπω θα εξυπηρετούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπω θα σα εξυπηρετούσε και εσά και εμά να φτάσουμε σε συμφωνία κάποια διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν ε, τεχνικοί φραγμοί στο να υλοποιηθούν αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν γίνει ένα τρίτο κράτος από την 1η Νοεμβρίου το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα είναι πλέον μέλος διαφόρων διεθνών οργανισμών όπως του Βορείου Ατλαντικού ή της προστασίας του τόνου ή άλλων οργανισμών. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε μήπως με κάποιες διασφαλίσεις αποφύγουμε τις ε, δυσκολίες και τα αδιέξοδα. Μήπως αυτό συμφωνήσει και η Βρετανική κυβέρνηση. Και μήπως υπάρχουν και άλλοι τεχνικοί φραγμοί, τους οποίους δεν έχουμε συζητήσει ακόμα. Ωραία. Μια ακόμα ερώτηση και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Γιατί και άλλοι έχουν ζητήσει τον λόγο βεβαίως. Θα τον δώσουμε. Ο κύριος Ρέισεν. Μάλλον το έχω προφέρει λάθος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για τις προτάσεις της. Μπορούμε έτσι να σκεφτούμε όλα τα πιθανά σενάρια, ό,τι μπορεί να προκύψει, ιδίω αν έχουμε ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Η συμφωνία, όπως είπαμε, θα προκαλέσει μόνο απώλειες και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει αποκλεισμένο στην ίσο της Βρετανίας, πράγμα που δεν βρίσκω να είναι θετικό ούτε για τους ίδιους, και ε, δεν είναι εύκολο φαίνεται να καταλήξουμε σε συμφωνία που να είναι υποφελής για όλους. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να προβλέψουμε και μέτρα κατεπίουσα ανάγκη εφόσον χρειαστεί, κυρίω τεχνικέ διευθετήσει. Διότι υπάρχουν ανησυχίε ιδίω για αυτό που ε, ακούστηκε και προηγουμένω, την αμεβαιότητα. Για του Ολλανδού αλληλεί, το σημαντικό είναι να ξέρουν αν από την 1η Νοεμβρίου και μετά θα μπορούν να αλλιεύουν στα Βρετανικά ύδατα ή όχι. Με τον κανονισμό αυτό έχουμε την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν ακόμα κανόνε. Κανόνε για τα για τα παραγαδιάρικα και εκεί χρειάζονται άδειε από τι Βρετανικέ Αρχέ για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να αναλάβουμε μέτρα από τη δική μα πλευρά μόνον, χωρί να ξέρουμε πώ αντιδρά το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να υπάρξει και από εκεί μια απάντηση. Πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε το θέμα τη αμοιβαιότητα για να δούμε αν θα μπορούμε να ψαρεύουμε αμοιβαίω στα είδα τα ημέν των δε. Πρόταση παράτασης της ισχύω των σημερινών κανόνων, λοιπόν, μέχρι το 2021, ίσως, αλλά γιατί όχι και μεγαλύτερη ισχύ. Ε, μπορεί να χρειαστεί και να συζητηθεί σύντομα. Ευχαριστούμε. Μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ακούσατε πολλά για την αμοιβαιότητα και την επιθυμία των αλλιέων, των ψαράδων, να ξέρουν λίγο σαφέστερα τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε ακριβώ βέβαια ακριβώς ποιο πλαίσιο θα δημιουργηθεί και θα προκύψει για να υπάρχει βιώσιμη αλεία για όλε τι πλευρέ τη παρατηρήση σα. Όμω ακούστηκε ότι η Βρετανική Αρχή πρόκειται να συμπεριλάβει στη δική τη νομοθεσία πολλέ από τι αρχέ τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Όμω, ε, λόγω ε, τη πάυση λειτουργία του Κοινοβουλίου, αυτή η συμφωνία και αυτή η προοπτική δεν ισχύει πλέον. Τι συμβουλέ θα δίνατε λοιπόν στου ψαράδε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για την τελευταία σας ερώτηση. Πολύ ενθαρρυντική και απλή. Πριν περάσω στις διάφορες παρατηρήσεις με λεπτομερείς κάποια δικά μου σχόλια. Είπα προηγουμένως ότι κάποια στιγμή η Βρετανική κυβέρνηση είχε πει ότι απλώς θα αντιγράψει στη μεταβατική περίοδο αρχές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, στη δική της, τη Βρετανική Νομοθεσία. Οπότε τα κοιτάζαμε μαζί. Για να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε την νομοθεσία τους στο μέλλον. Το είχαν πει προηγουμένως βέβαια. Αλλά είπα επίσης ότι δεν υπάρχει πια καμιά βεβαιότητα ότι αυτό θα συμβεί βάσει των σημερινών στοιχείων. Για την αμοιβαιότητα. Ίσως δεν ήμουν αρκετά σαφής. Δεν προκύπτει εδώ αμοιβαιότητα, δεν προκύπτουν ούτε προσδοκίε περί αμοιβαιότητα. Αυτό που θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αν κάποια στιγμή υπάρξει αμοιβαιότητα, βραχυπρόθεσμα μετά από ένα σκληρό Brexit, τεχνικώ θα είμαστε πλήρω προετοιμασμένοι. Δεν έχει σκοπό η πρόταση αυτή να είναι σημείο αφετηρία για διαπραγματεύσει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε ότι η γραμμή τη Ένωση εφόσον περατωθεί η διαδικασία χώρισε από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι να μην έχουμε εν μέρη αποσπασματικέ συμφωνίε στον ένα ή τον άλλο τομέα ή χώρο πολιτική. Η συμφωνία περιεμβεβαιότητα περι θα προκύψει στο μέλλον, εάν προκύψει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο άλλωστε με νομοθετικέ προτάσει. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε λοιπόν την αμοιβαιότητα και εξ αυτού υπάρχει ένας τεράστιος βαθμός ανασφάλειας που δεν μπορεί να την απαλύνει ούτε αυτή η πρόταση ούτε κάτι άλλο μελλοντικά για το ποια θα είναι η κατάσταση ως προς την πρόσβαση από την 1η Νοεμβρίου. Αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε αργότερα. Δυστυχώ δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι κανεί σε θέση να μαντέψει τι θα συμβεί. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναρξη διπραγματεύσεων ή το να δημιουργήσουμε προσδοκίε περί αμοιβαιότητα. Όπως είπε και ο συνάδελφός μου και υπενήχθηκε, Το θέμα είναι ότι ε, έτσι κι αλλιώς εδώ έχουμε μια μονομερή αντίδραση. Εμείς κοιτάζουμε να προετοιμαστούμε για το μελλοντικά ενδεχόμενα. Η Βρετανική πλευρά θα δούμε αν έχει προετοιμαστεί για να απαντήσει αναλόγω. Πάντω αυτή είναι η προετοιμασία η δική μα εφόσον προκύψει η κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Δεν ανοίγουμε διαπραγματεύσει. Αυτό είναι το πρώτο νομίζω που ρωτήσατε. Και επίση είναι αλήθεια ότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει χωρί συμφωνία την 1η Νοεμβρίου, θα είναι πραγματικά ένα ανεξάρτητο τρίτο παράκτιο κράτο και θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλο του διεθνού οργανισμού. Δεν είναι δική μα ευθύνη αυτό. Εμεί είμαστε ούτω ή άλλω μέλη. Και γνωρίζουμε από την επίσημη επικοινωνία μα ότι είναι προετοιμασμένοι για μια τέτοια προοπτική. Οι βασικοί οργανισμοί και οι σχετικέ αιτήσει ήδη εξετάζονται. Αλλά είπατε εσεί για του φραγμού, τα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν. Αυτό είναι ένα από αυτά. Εφόσον υπάρξει σκληρό Brexit. Οπωσδήποτε ισχύει. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει την ευθύνη. Ευθύνη όχι μόνο για τα δικά του τα συμφέροντα, αλλά γενικώ να διασφαλίσει ότι θα πρέπει να έχει συμμετοχή εκεί που πρέπει να έχει συμμετοχή θα πρέπει να κάνει αίτηση για να γίνει μέλος. Οι περισσότεροι οργανισμοί είναι έτοιμοι να εξετάσουν τέτοιου είδου αιτήσει. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα να ακολουθήσουν αυτή την οδό. Τώρα, άλλη τεχνική φραγμή. Στι διαπραγματεύσει μα τα τελευταία τρία χρόνια και στη δική μα προετοιμασία για ένα σχέδιο έκτακτη ανάγκη, το τελευταίο χρόνο, Χρειάστηκε να δούμε όλες τις τεχνικές ελλείψεις και τα εμπόδια. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας. Αυτά θέλαμε να διασφαλίσουμε κυρίως. Εκπλήξει υπάρχουν πάντοτε. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι είμαστε καλά προετοιμασμένοι για το οποιοδήποτε από τα ενδεχόμενα μπορεί να προκύψουν. Και για τα σημεία εδώ και τρία που ανέφερε και ο Πρόεδρος. Είμαστε έτοιμοι και για τις τρεις αυτές προοπτικές. Δεν νομίζω ότι από τη δική πλευρά υπάρχουν άλλα τεχνικά κολλήματα. Τώρα από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου μετά για τις ε, ανταλλαγές, τα swaps δεν πρόκειται να το αρνηθούμε αυτό και για τις ανησυχίες των ψαράδων και της βιομηχανίας έχουμε επιτρέψει μια μεταβατική περίοδο, σε μια πρώτη φάση, να συνεχιστεί το σύστημα των ανταλλαγών. Είναι σημαντικό αυτό για τη μικροδιαχείριση τη αλληλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετησίω περίπου 2.000 ανταλλαγέ ποσοστώσεων ε, προκύπτουν μεταξύ των κρατών μελών. Διευκολύνει αυτή τη δουλειά των ψαράδων. Εάν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, νομίζω 30-40% ε, των δυνατοτήτων ανταλλαγή θα καταρρεύσει. Και η αλληλευτική βιομηχανία και τα κρατημέλη έχουν εκφράσει σοβαρέ ανησυχίε για την ε, απώλεια μιας τέτοιας δυνατότητας και για τις ε, παρενέργειες που μπορεί να έχει στην καθημερινή μικροδιαχείριση της αλληλευτικής δράσης. Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι ποσοστώσει θα συνεχίσουν καθημερινά να μπορούν να ανταλλάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω και η όλη πρότασή μα για την κατάσταση εκτακτή ανάγκη έχει μονοετή διάρκεια και θα πρέπει να δούμε τι θα προκύψει στο μέλλον και πώς θα διαμορφωθεί το σύστημα ανταλλαγή ποσοστώσεων. Πάντως είναι μια απέτηση της πραγματικότητας και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Η πρόταση της Επιτροπής και της Ένωσης είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε και προβλεπόταν μόνο για το 19 στην αρχή της ε, όλης δουλειάς μας. Τώρα κάναμε πρόταση και για το 2020 εφόσον προκύψει το ενδεχόμενο του Brexit χωρίς συμφωνία. Περιορισμένη λοιπόν διάρκεια, αναγκαστικά αυτοπεριοριστήκαμε. Νομίζω ότι απέντησα τις περισσότερες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Διεξοδική απάντηση. Η βασική ερώτηση είναι ότι ο κάθε ψαράς, ασχέτως εθνικότητας, θέλει κάποια ασφάλεια. Αυτό ήταν και το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων που κρατάνε εδώ και τρία χρόνια. Και πέντε, εδώ και πέντε εβδομάδες ή όχι λέτε, κανείς δεν είναι σε θέση να κρίνει το τι θα συμβεί το Νοέμβριο. Πέντε εβδομάδες μείνανε μετά από τρία χρόνια διαπραγματεύσεις και ψαράδες και πάλι, εμείς και πάλι, δεν ξέρουμε τίποτα. Έτσι είναι, έτσι. Ο κύριος Μηγιανμόν. Ναι και όχι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Ούτε κανείς να προβλέψει με ασφάλεια που θα είμαστε την 1η Νοεμβρίου αλλά να είμαστε και ρεαλιστέ. Έχουμε εξαντλήσει όλες τις διαφορετικές δυνατότητες, τι έχουμε κοιτάξει όλες. Ε, συμφωνή, απουσία συμφωνίας. Θα το συζητήσουμε και αυτό μετά. Μπορεί να υπάρξει Brexit χωρίς συμφωνία. Δύο εναλλακτικές προκύπτουν εδώ. Πρώτα απ' όλα, όντω να μην έχουμε πρόσβαση στα βρετανικά ύδατα, οπότε χιλιάδε ε, Ευρωπαίων ψαράδων θα έχουν ε, μεν σαφήνεια του τι συμβαίνει, αλλά πολύ αρνητική εικόνα. Δεν είναι λοιπόν ε, ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα διαφορετικά σενάρια. Και το τρίτο είναι αυτό που λέμε τώρα. Brexit χωρί συμφωνία, όπου το, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο ανοίγει τα ύδατα του του Ευρωπαίου τουλάχιστον ψαράδε για ένα διάστημα. Και υπάρχει εδώ αμοιβαιότητα και αυτή είναι μια κατάσταση σαφήνειας. Αλλά και εκεί θα πρέπει να δούμε τις τεχνικές λεπτομέρειες και γι' αυτό τις κοιτάζουμε. Δεν λέω ότι, ξεκινά, ότι ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά δεν ξεκινάμε και από το μηδέν. Έχουμε κοιτάξει με λεπτομέρεια τα διαφορετικά σενάρια που μπορεί να προκύψουν και όλα ανησυχούν, αλλά κάποια είναι κάπως καλύτερα από τα άλλα. Προφανώ προτιμάμε να υπάρξει Brexit χωρί συμφωνία, αλλά με μεταβατική περίοδο, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα Βρετανικά τα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα ήταν πολύ καλύτερο σε μια αφετηρία για όλου. Όταν ξυπνήσουμε το πρωί τη 1η Νοεμβρίου. Αλλά έχουμε χαρτογραφήσει όλα τα διαφορετικά σενάρια. Ευχαριστώ. Μα αρέσει πολύ αυτή η, η, η έννοια τη αρνητική αφήνεια. Να πούμε τώρα ότι συζητάμε για τα σημεία 4 και 5 του σέλος αυτό αυτά τα 2 και 3 τα απομακρύναμε. Σημαντικό θέμα. Πολύ καλά κάνατε. Και συσχετίσατε τα δύο σημεία της μερίσιας διάταξης. Και στην Ολομέλη στο Στρασβούργου πριν από λίγες μέρες το συζητήσαμε. Και πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν στο έγγραφο σε σχέση με το έγγραφο Hammer. Και πραγματικά υπήρχε το ενδεχόμενο ε, να υπάρξουν επεισόδια μεταξύ Ευρωπαίων και Βρετανών αλλιέων. Αν υπάρξει Brexit χωρίς συμφωνία και χωρίς πρόσβαση στα ύδατα, είναι πολύ δύσκολο θέμα. Και σίγουρα υπάρχουν άλλες προοπτικές ε, και γινόταν λόγος μέχρι και για βία, βίες ενέργειες. συμφωνούμε νομίζω περισσότερο ότι θέλουμε να υπάρχει ε, συνέχιση των σχέσεων με τον Ομένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά τα είδα, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα και υπάρχουν αυτά τα έκτακτα τεχνικά μέτρα που βέβαια πρώτα θα πρέπει να εγκριθούν και από τις δύο πλευρές πρωτού εφαρμοστούν στην πράξη. Αλλά αν υπάρχει αυτή η συμφωνία αμοιβαίας πρόσβασης, πρέπει να είμαστε τεχνικά έτοιμοι και θα πρέπει να υπάρξουν και οι σχετικές τροποποίησεις στον κανονισμό. Σε ό,τι αφορά τώρα το μέλλον, θα έχουμε μια πολυδιάστατη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ένα θέμα που είναι προτεραιότητα για την Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο. Είναι η Γαλλία που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των σχέσεων των δύο πλευρών Υπάρχουν και κάποιοι που αποκλίνουν και διαφωνούν, αλλά τι γίνεται με την αλληλευτική και την εξωτερική δραστηριότητα. Είναι θέμα πρόσβαση στην αγορά των προϊόντων των αλληλευτικών και εδώ μιλάμε για την πρόσβαση στην αγορά της υπηρετικής Ευρώπης. Υπάρχουν πρώτα αλληλευτικά τα οποία εξάγουν οι Βρετανοί στην ε, υπηρετική Ευρώπη και αντίστροφα. Πάντοτε η προσέγγιση πρέπει να ακολουθήσουμε πρέπει να είναι συνολική, να μην βλέπουμε μόνο την εξωτερική δραστηριότητα, πρόσβαση σε πόρου, και, αλλά να, δεν βλέπουμε και την πρόσβαση στις αγορές. Για να είναι πιο ισορροπημένη σχέση με αυτόν τον τρόπο. Και στο μέλλον, σε αυτή τη μακροσυμφωνία μιας μεγάλης οικονομικής εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένου Βασιλείου που όλοι επιθυμούμε, αν γίνει Brexit τελικά, αυτή η οικονομική συμφωνία, αυτή η μεγάλη οικονομική εταιρική σχέση θα πρέπει να συνοδεύεται κατά ανάγκη και από μια συμφωνία για πρόσβαση σε ύδατα και πόρους. Δεν μπορώ να φανταστώ μια μελλοντική σχέση με τον Ηνωμένο Βασίλειο που η Ένωση δεν θα έχει πρόσβαση σε πόρους και ύδατα. Άρα μεγάλη οικονομική εταιρική σχέση και συμφωνία αμοιβαία για την πρόσβαση σε πόρους και ύδατα πρέπει να πάνε από κοινού αυτά τα κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Η συνάδελφος από το κόμμα του Brexit λέει ότι ανησυχούν πολύ στην αίθουσα. Βεβαίω και ανησυχούμε. Και ανησυχούμε όταν εγώ άκουσα κάποιοι να μιλάνε για τον Brexit, είπαν ότι εμεί θα πάρουμε τον έλεγχο των υδάτων μα η Βρετανία λύση, θα κάνουν ό,τι θέλουν στα νερά τους χωρίς να σκέφτονται τίποτα και θα αλλιεύουν ό,τι θέλουν. Φυσικά και ανησυχούμε λοιπόν με αυτά. Γιατί αύριο μπορεί να γίνεται ό,τι να είναι στα βρετανικά είδατε, Αλλά τα ψάρια δεν ξέρουν ε, από σύνορα και από αποκλειστικέ οικονομικές ζώνες, άρα ό,τι γίνεται στα βρετανικά ύδατα μας αφορά. Όπως και να έχει, είμαστε σε μια περίοδο που θέλουμε να εφαρμόσουμε την κοινή ελευθερική πολιτική. Αν δείτε τι γίνεται στην Βόρεια Θάλασσα, στη στον Ατλαντικό ε, και στη, προς τη Σκοτία, γίνονται προσπάθειες από τους Αλίσσα, υπάρχουν ελευτικές προσπάθειες από τους Ευρωπαίους, από τους Βρετανούς ψαράδες και όλα αυτά θα τα θέσουν από αμφισβήτηση, όπου η βιωσιμότητα των πόρων θα ξανατεθεί ε, υποσυζήτηση. Φυσικά και ανησυχούμε όταν ακούμε τη Βρετανική κυβέρνηση να μιλάει για την αμοιβαιότητα. Που είναι αυτό που ξανανοίγει σήμερα. Ο Μάικλ Γκόβ όταν ε, ήταν υπεύθυνο για το περιβάλλον, υπουργό έλεγε ότι θα υπάρξει πρόσβαση στα Βρετανικά για τους αλλιευτικούς ε, για τους Ευρωπαίους αλλιείς. Αυτό το είπε στη συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων. Δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη τέτοια δήλωση. Μα ανησυχεί λοιπόν το Μεσαλία, αλλά μας ανησυχεί και το θέμα της βιωσιμότητα των πόρων. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, για ποιο λόγο τα μέλη του κόμματο Brexit συμμετέχουν και παρεμβαίνουν στη συζήτηση αυτή. Τι τους νοιάζει τα γίνοντα τον Brexit. Εσείς κάνατε την καμπάνια σα να φύγετε από την Ένωση, κάνατε καμπάνια υπέρ του Brexit. Εσείς μας λέτε, εσείς οι εκπρόσωποι των εκλογέων, των ψηφοφόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην αναμειγνύεστε πλέον στα εσωτερικά μας. Mind your business, θα θέλω να σας πω κι εγώ. Mind your own business, λοιπόν. Αυτό θέλω να σας πω κι εγώ. Τα δικά σας να κοιτάτε, τη, δουλειά σας. Η κυρία Dodds, η κυρία Ντότζ έχει το λόγο, λέει ο Πρόεδρο. Uh, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Όπως τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η τεράστια πλειοψηφία των αλλιευτικών κοινοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε υπέρ της αποχώρησης. Και αυτό διότι αντιλαμβάνεται ότι η διαδικασία μέσω της οποίας υποχρεωνόταν να αλλιεύσει ήταν άδικη και κατά των συμφερόντων της. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε το γεγονός αυτό κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής και σε οποιαδήποτε περίπτωση τέλος Οκτωβρίου ή όχι το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτο κράτος και θα αναλάβει την αποκλειστική διαχείριση και εκμετάλλευση των υδάτων του. Τώρα εγώ έχω πολλά χρόνια εμπειρία στην Επιτροπή αυτήν να συζητούμε για την πρόσβαση σε βρετανικά υδατά. Έχω συναντηθεί με πολλούς αλληλείς που λένε ότι το 60% των εκφορτώσεών τους προέρχεται από τη Βόρεια Θάλασσα. Το 90% του συνόλου του γάδου είναι στα στενά που αλλιεύεται. Και γι' αυτό αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια αντίληψη άδικης μεταχείρισης. Άδικης μεταχείρισης από πλευρά των, Βρετανιών, των Βρετανών αλλιέων. Και κάτι που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Οι Βρετανοί αλλιείς προχώρησαν σε αποφασιστικά βήματα για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της αλλιευτικής τους ε, δραστηριότητας. Όταν εγώ πρώτο έγινα μέλος της Επιτροπής αυτής, η ρέγγα της Ιρλανδικής θάλασσας ήταν υπο... σε κίνδυνο και σήμερα είναι βιώσιμο απόθεμα. Αυτό είναι απόδειξη της ε, υπεύθυνης τάσης που τήρησαν οι Βρετανοί αλληλείς. Και το Brexit δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Το έχουν κατανοήσει και έχουν αναλάβει πολύ υπεύθυνα και αποτελεσματικά μέτρα. Ακούσαμε πολλά σήμερα στη συζήτηση για την αμοιβαιότητα. Εκτιμώ απολύτω τη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η τροποποίηση αυτή, η τροπολογία αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει μια προσδοκία αμοιβαιότητα γιατί εξαρτάται από τη διαπραγμάτευση των δύο πλευρών. Αλλά γενικώ συζητώντα για την αμοιβαιότητα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στο πώς χρησιμοποιούμε τους όρους. Στις 18 Σεπτεμβρίου μια αξιόπιστη Ιρλανδική εφημερίδα δημοσίευσε τη δήλωση μιας πολύ μεγάλης αλλιευτικής οργάνωσης σχετικά με αντιπαραθέσεις στη θάλασσα ε, ε, στα ανοιχτά της ακτής. Ε, αναφέρεται χάος και συγκρούσεις στη θάλασσα, αποκλεισμοί, εμπάργκο και ιδιαίτερα προβλήματα στην Ιρλανδική θάλασσα, στα βορειοδυτικά του Ντόνεγκαλ και στα στενά της Μάνχης και στη Βόρεια θάλασσα. Αναφέρθηκαν και δυνητικά βία περιστατικά Είχαμε πει, πάρει μια γεύση πέρυσι με την ε, αντιπαράθεση που είχαμε σχετικά με αντιλαμβάνεται, εν πάση το Ηνωμένο Βασίλειο πόσο σημαντική είναι η προσβασιμότητα στα ύδατα ε, ε, και συνολικά για τις βόρειες θάλασσες της Ευρώπης. Εδώ είμαστε νομοθέτες. Ε, δεν είμαστε παραβάτες. Τηρούμε τον νόμο, δεν τον παραβιάζουμε. Η Επιτροπή αυτή λοιπόν είμαι σίγουρη ότι τέτοιου είδους ορολογία όπως αυτή που δημοσιεύτηκε στις 18 Σεπτεμβρίου θα καυτηριαστεί. Αυτό δεν βοηθά κανέναν. Εγώ πολύ λυπούμε που τέτοια άρθρα δημοσιεύονται, που χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα, αλλά δεν μπορούμε να υποκύπτουμε και σε απειλές βίας ή εμπλοκών ή αντιπαραθέσεων. Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι και εσείς θα το καταδικάζετε αυτό και θα συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν είναι ο τρόπος για να προχωρήσουμε. Οι διαπραγματεύσεις που είχαμε για το Σκουμπρί, για παράδειγμα με την Ορβηγία και άλλους, δεν χρησιμοποιούν τέτοια ορολογία. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, που μακρηγόρησα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι, όλα τα μέλη εκτιμούν τα σχολεία της σας. Η ε, κυρία Σάλιβαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πράγματι βρισκόμαστε σε αβέβαιους ε, καιρούς και κατόπιν και των σχολείων κάποιων άλλων ομιλητών μετά το τέλος Οκτωβρίου θα υπάρξει μια χαοτική κατάσταση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και μετά και την έκθεση Yellow Hammer στο Ηνωμένο Βασίλειο. όπου αναφέρεται και η δυνατότητα παράνομης αλίευσης των Ευρωπαίων αλίεων στα Βρετανικά ύδατα. Τι κάνει η Επιτροπή έχει μιλήσει με τα κράτη-μέλη προκειμένου να αποτρέψει περιστατικά συμπλοκές Τι μπορούμε να κάνουμε για την αμοιβαία δυνατότητα πρόσβασης για να προστατεύσουμε τις αλληλείς και για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοια περιστατικά στη θάλασσα. Thank you, ευχαριστώ Πρόεδρε. Διαδικαστικά, επειδή είπατε ότι συζητούμε και για το 5, θα περίμενα να έχουμε μια εισαγωγή από πλευρά του εκπροσώπου της Κομισιόν. Και τουλάχιστον να χρησιμοποιήσουμε την εισαγωγή του, μια και σίγουρα θα έχει προετοιμαστεί γι' αυτό, για να υποβάλουμε ερωτήματα. Τώρα, η αμοιβαία πρόσβαση και η προετοιμασία της, αλλά χωρίς να την έχουμε την ίδια την αμοιβαιότητα, είναι λίγο προβληματική κατάσταση, γιατί ε, το να έχει κανείς, το να εξασφαλίσει αμοιβαιότητα δεν υπέφτει από τον ουρανό, απαιτεί σοβαρή δουλειά, σοβαρή προετοιμασία. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις μας εξηγείται ότι ο κανονισμός για τις επιταχυμένες διαδικασίες ώστε οι, ευρωπαϊκοί, οι Ευρωπαίοι αλληλείς να έχουν πρόσβαση στα Βρετανικά ύδατα θα λάβουν χώρα και θα επεκταθεί και η Βρετανική πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά ύδατα. Θα έχουμε λοιπόν fast tracking και από την ε, ευρωπαϊκή πλευρά ή μήπως θα έχουμε side tracking. Δηλαδή θα επιταχύνεται τη διαδικασία ή θα τοποθετήσετε εμπόδια. Ο κ. Βαντάλεν είπε ότι δεν θα υπάρξουν νικητές από τον Brexit. Δεν θα σας είναι έκπληξη ότι διαφωνώ με τη δήλωση αυτή και ένα παράδειγμα θα ήταν ότι θα μπορούσαμε να σταματήσουμε στα Βρετανικά ύδατα απαράδεκτες αλλιευτικές ε, πρακτικές που αυτή τη στιγμή επιτρέπονται. υπάρχουν διάφορα μέτρα που θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρξει οποιαδήποτε αμοιβαιότητα στα θέματα ε, πρόσβασης στα ύδατα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θέλουν να κάνουν ερωτήσει, αλλά πριν παραγίνει μακρύ ο κατάλογο, ίσως η Κομισιόν να, να δώσει κάποιες απαντήσει τώρα. Θέλουμε να αποφύγουμε συγκρούσεις και αντιπαραθέσει. Αυτό είναι ο στόχο. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε τι συζητήσεις έχουν γίνει μεταξύ Ηνωμένου Βασίλειου και Ένωση για να μην υπάρξουν τέτοιε συγκρούσει. και επειδή συζητείτε το θέμα του ότι μπορεί να εκδιωχθούν υποορισμένε περιστάσεις από τα βρετανικά ε, χωρικά έδατα, τα ληφτικά σκάφη της θα γίνει και το ανάποδο. Και αυτό που είπε ο κύριος Μόντι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μήπως θα μπορούσατε να κάνετε μια εισαγωγή Ευχαριστώ και εγώ. Βλέπω ότι προχωρούμε, έχουμε μετακινηθεί σε ευρύτερα σενάρια και υποθέσεις και δεν περιοριζόμαστε στη συζήτηση του συγκεκριμένου μόνο σημείου της ημερήσιας διάταξης. Ο Ισπανός που μίλησε να επιβεβαιώσω ότι ναι, ε, θα, είμαστε, ε, θα έχουμε ως βάση τις κατευθύνσεις γραμμές του Συμβουλίου στην περαιτέρω εργασία μου. Και χαίρομαι που εκτιμά την πρόταση. Καλό είναι αυτό. Για το χάος και το ενδεχόμενο συγκρούσεων, αντιπαραθέσεων. Να πω τι κάνουμε πέραν της πρότασης αυτής τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε πολύ στενές επαφές με τα οκτώ κράτη μέλη που έχουν αλλιευτικά δικαιώματα σε, μέρη των, σε τμήματα χωρικών υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου άλλα, για άλλα κράτη νησιού όπως η Φιλανδία για παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν τα οκτώ βασικά κράτη. Έχουμε συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να συντονίσουμε την αντίδραση των κρατών μελών στα διάφορα πιθανά σενάρια και περιλαμβάνεται εδώ και η αποφυγή συγκρούσεων. Εκ μέρους όλων των κρατών μελών μπορώ να πω ότι όλα τα κρατημέρια αντιλαμβάνονται το ενδεχόμενο να υπάρχουν αντιπαραθέσεις αν είναι κλειστά στα ευρωπαϊκά σκάφη τα βρετανικά χωρικά ύδατα, μάλλον τα βρετανικά λευτικά ύδατα. και προετοιμάζονται στις στρατηγικέ του τα κράτη-μέλη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και εμεί προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έλεγχου της που δραστηριοποιείται και συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για στρατηγικέ ελέγχου και για τον εντοπισμό παράνομη άναρξη αδέλου της Αλίας γιατί πέφτουμε πλέον και εδώ. Γιατί θα τον αντιμετωπίζουμε ως τρίτο εταίρο, διεθνή εταίρο του Ηνωμένου Βασίλειου. Αν υπάρξει χάος, ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, υπάρχει το ενδεχόμενο για αντιπαράθεση, για σύγκρουση, αλλά εργαζόμαστε σκληρά ώστε να το αποφύγουμε το ενδεχόμενο αυτό ή να το περιορίσουμε στο ελάχιστο. Βέβαια όλα είναι απρόβλεπτα, αστάθμητα, γιατί πρόκειται για κάτι εντελώς ε, καινοφανές, πρωτόγνωρο. Ίσως όμως θα αντιμετωπίσουμε ε, παρά την προετοιμασία μας απρόβλεπτα φαινόμενα. Εξίσου σημαντικό είναι ότι επικοινωνούμε απευθείας με τους εμπλεκομένους φορείς, ελευτικές ενώσεις κύριους και άλλους και τους αναφέρουμε και τις ευθύνες τους βέβαια, αλλά ξεκαθαρίζουμε και κάποιες καταστάσεις. Έχουμε ένα σημείωμα για αυτούς τους ε, ενδιαφερομένους δεν ξέρω, ήδη από τον Αύγουστο-Ιούλιο του 2018 και πρόσφατα τον Ιούλιο του 2019 δημοσιεύσαμε ένα μακρύ κατάλογο απαντήσεων που δίνουν πολύ πρακτικές οδηγίες στους αλλοίς και όχι μόνο και στις αρχές διαχείρισης. Άρα, προσπαθούμε να προετοιμαστούμε από κοινού με τους εμπλεκομένους για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. παρόδου. Για το σχόλιο της κυρίας Ντότς, μια μικρή διόρθωση για την ε, διαχείριση της ρέγκας ε, στο Ελλαδικό Πέλαγος. Κοιτάξτε, ναι, πράγματι υπάρχει αλλά η προσπάθεια της Ένωσης είναι να είναι ε, βιώσιμη η αλία αυτού του είδους και όχι τόσο βρετανική προσπάθεια, πιο πολύ ενωσιακή. Ένας από τους τελευταίους ομιλητές μίλησε για την ταχεία διαδικασία, για την έγκριση αδειών. Κοιτάξτε, στέλνουμε έτοιμα ε, στο νομοσύλιο και έχουμε την ταχεία διαδικασία. Αν θα στέλνουν αντίστοιχα αιτήματα, δηλαδή να ψαρεύουν αλίστους στα δικά μας έτατα, θα έχουμε πάλι ταχεία διαδικασία. Εμείς προετοιμαζόμαστε από πλευράς μας. Αλλά καλό ήταν να υπάρξει και συνεργασία. Δεν θα μιλήσω για τις μηχανότρατες ε, με τα σειρώμενα. Θα δούμε. Ε, ε, θα δούμε. γιατί στόχος μας είναι να διατηρηθούν τα αποθέματα. Άρα όλοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να ξέρουν τι δικαιώματα έχουν, αλλά και τι υποχρεώσεις. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Δεν ξέρω μήπως μου ξέφυγε τίποτε. Αυτά έχω γράψει πάντως. Ο κ. Μιγιαμόν, λέει ο πρόεδρος, είπε για το ότι πολλά ψάρια από το Ηνωμένο Βασίλειο καταλήγουν ε, στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Και αν δεν υπάρχει πρόσβαση, δεν θα έχουμε στοιχεία ημερολογίου πλοίου. Ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Πώς θα βοηθήσει αυτό τη ρύθμιση μη της αλίας. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, όλες ε, οι μεθορικές ε, διατάξεις που ισχύουν ε, για τρίτα κράτη θα ισχύει το Ηνωμένο Βασίλειο. Έλεγχοι στα σύνορα, έλεγχος της άναρχης αηλίας και τα λοιπά, γιατί γίνεται τρίτη χώρα το Ηνωμένο Βασίλειο που πρέπει να τηρεί την νομοθεσία IUU. Αυτά είναι τα βασικά. Τις λεπτομέρειες μπορούν να σας πούν ειδικοί. Και φυσικά μας ενδιαφέρει ότι εξαρτάται πολύ από την αγορά της Ένωσης ε, η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, για την ε, πορεία των προϊόντων της. Άρα θα το έχουμε και αυτό υπόψη όταν ξεκινήσουμε τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και ξέχασα τι μου με ρωτήσατε. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα διάφορα σενάρια. Αν έχουμε συμφωνία αποχώρηση που θα την εγκρίνουν και οι δύο πλευρές και είμαστε σε μεταβατική περίοδο, τότε η βάση μας είναι συνεργατική διαχείριση. Θα τηρεί δηλαδή την κοινελευτική πολιτική των Ηνωμένων θα συμμετέχει και θα τηρεί τους κανόνες, άρα θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Αν όμως έχουμε σκληρό Brexit χωρίς συμφωνία από το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να μην χορηγήσει πρόσβαση στα έδατά του και εμείς αποφασίσουμε να μην χορηγήσουμε πρόσβαση στα έδατά μας, δεν θα έχουμε τόσο συνεργατικό κλίμα και περιβάλλον. Άρα πρέπει υπό το πρίσμα του κάθε σενάριου να δούμε τα πράγματα και να προβλέψουμε τι θα γίνει από τότε. Αν χωρίσουν οι δρόμοι μας ε, όχι φιλικά, τότε θα δούμε πώς θα ρυθμίσουμε. Γιατί όλα τα στοιχεία είναι αντικείμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων για τη συνεργασία και τη συνδιαχείριση. Αλλά αν έχουμε σκληρό Brexit και κλειστά έδατα με κατέρωθεν, φυσικά η συνεργασία θα είναι πολύ μικρή. αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα προκύψει και αν θέλουν και πόσο γρήγορα θέλουν να αποκαταστήσουν τα πράγματα δύο πλευρές. Αλλά ναι, αλήθεια είναι. Έχουμε κοινά αποθέματα, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Τι θα γίνει με τον έλεγχο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και για το μέλλον το θέμα του ελέγχου. Αυτό το σχόλιο δεν αφορά τις διαπραγματεύσεις. Λόγω των πόρων απαιτείται να δίνετε συνεχής προσοχή. Κυρία Μπιλμπάου, καλημέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο συγγνώμη, αλλά ήμουν στην Επιτροπή Μεταφορών που είχαμε ψηφοφορίες και δεν ήμουν από την αρχή. Όμως είναι προφανές να άκουσα ότι υπάρχει πρόδειλη ανησυχία έναντι ενό Brexit σκληρού χωρί συμφωνία. Μιλήσαμε για, κα, για χάο, για συγκρούσει στη θάλασσα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε αυτά να τα αποφύγουμε και να μην συμβούν τέτοια φαινόμενα. Όπω ε, πάντα πράγματα όμω, ε, μέρα τη μέρα, υπάρχουν κάποιε υποθέσει που διαμορφώνονται. Μία υπόθεση είναι μόνη τροποποίηση που, που ενοχλεί είναι οι συμφωνίες της Μεγάλης Παρασκευής. Και όταν μιλάμε για την παραθέση πρώτες τέτοιες συγκρούσεις θα μπορούσαν να είναι στα σύνορα που θα υψωθούν μεταξύ των δύο τμήματων της Τριλανδίας. Πάω πιο πέρα όμως. Οι πληγήσεις χώρες, οι θυγόμενες, είναι οκτώ είπατε, οκτώ κράτη-μέλη. Πέραν του ελέγχου, του συντονισμού, Σίγουρα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά. Ρωτώ την Επιτροπή. Ξέρει ή γνωρίζει ή πιστεύει ότι εργάζονται τα κράτη-μέλη ε, με βάση τη χειρότερη υπόθεση, δηλαδή του Brexit χωρίς συμφωνία, όπου ένα μεγάλο μέρος του στόλου θα μπορούσε να μην έχει πλέον αλληλευτικές δυνατότητες. Πέραν των μέτρων ελέγχου. Προβλέπεται ε, να υπάρξει κάποια είδου βοήθεια, διατυπώνεται κάποιες προτάσεις ώστε ο κλάδος να μπορεί να αναδιαρθρωθεί, να αποκτασταθεί, να επιβιώσει, να σκεφτεί το μέλλον του. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Και δεύτερο, και άλλη μελλοντική υπόθεση και αυτή. Φυσικά. Σκοτία, αν υπάρξει τέτοιο ε, Brexit, χωρίς συμφωνία, σκληρό Brexit, ανακοινώνει ήδη τη διεξαγωγή δημοψηφίων. όπου θα τίθεται και το ερώτημα αν θέλουν να είναι μέλη της Ένωσης. Μια τέτοια υπόθεση τι αλλάζει σε αλληλευτικές συμφωνίες, αν η Σκοτία ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ίσως ε, νωρίς για ένα τέτοιο ερώτημα, αλλά υπάρχουν και τέτοια σενάρια. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό θα άλλαζε πολύ τα πράγματα. Γιατί η Σκωτία έχει αλληλευτικά δικαιώματα. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Έχω τρία μέλη που έχουν ήδη τοποθετηθεί και θέλουν κάτι πρόσθετο. Θα σας ζητήσω να είστε σύντομοι. Ο κύριος Γκονθάλες επίσης ζήτησε... Κλείνω τώρα τον κατάλογο, έτσι. Παρακαλώ. Ναι, είναι σαφές πρόεδρε ότι το Brexit είναι πρόβλημα και ότι η άτακτη αποχώρηση είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αυτή που έλαβε την απόφαση να εξέλθει από το νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Εγώ προέρχομαι από την γαλήθεια με σημαντικά σκάφη που ενέχονται στο θέμα της αμοιβαία πρόσβασης. Εμείς δεν επιθυμούμε άτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά βλέπουμε ότι μπορεί δυνητικά να δημιουργηθεί χαοτική κατάσταση. και σε μια περίπτωση άτακτης αποχώρησης με το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτο κράτος, τρίτη χώρα, θα πρέπει να είχαμε μια σταθερότητα, θα πρέπει να κατανείμουμε σωστά τα αποθέματα. Αν όμως το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει ατάκτος χωρίς να συμφωνήσει, αυτές οι πρακτικές που μέχρι τη στιγμή στηρούνται, ίσως να μην τηρούνται στο μέλλον. Τι θα γίνει λοιπόν σε μια τέτοια περίπτωση, θέλω να ρωτήσω την ε, Κομισιόν και να εκφράσω την ε, ανησυχία μας για το χάος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί και για στόλους που ε, λειτουργούν υπό Βρετανική σημαία, αλλά ε, ιδιοκτησίας μη Βρετανικής, λέει ο ο κύριος Αλάκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και την συνάδελφο που ανέφερε το, στη Σκοτία γιατί το μέλος της, ε, ε, ε, των υδάτων των σκοτσέζικων αλλά και εν γέννη της Σκοτίας εντός του προβλήματος του Brexit είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπε και ο κύριος Μόντιφ, πολύ ε, λυπούμε που δεν είχαμε μια εισήγηση της Κομισιόν για το σημείο 5. Ήταν σημαντικό γιατί πολλοί ανησυχούν. Ο συνολικός κλάδος και οι ελείς και οι μεταποιητές και τα μικρά σκάφη ε, σχετικά με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα είναι σημαντικό όχθο μετά την 1η Νοεμβρίου. Μιλούμε για 160 στερλίνες αναποστολή τέτοιου άκθους. Και τι θα γίνει με τη βιωσιμότητα των μικρών αλληλευτικών σκαφών αν έχουμε χαοτική και άτακτη αποχώρηση. Θα πρέπει να σταματήσουν για δύο ή τρεις εβδομάδες. Και αυτό σημαίνει μάλλον για πολλά από αυτά που θα χρειαστεί να αποσυρθούν, να σταματήσουν τη δραστηριότητά του. Και αυτό θα ισχύσει για του εξαγωγεί επίση. Οπότε ρωτώ, η σημερινή Βρετανική κυβέρνηση έχει ζητήσει ε, εξαίρεση από τις ε, παρούσες διατάσεις ε, υγειονομικών πιστοποιητικών. και αντιλαμβάνομαι και τα όσα λέμε σχετικά με την ε, ευθυγράμμιση που θα μπορούσε ή να, να, λάβει ή να μην λάβει χώρα από βρετανική πλευρά νομοθετικά. Έχετε κάνει δηλαδή κάποια δουλειά και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και με την σημερινή που θα μπορούσε να υλοποιηθεί άμεσα. Και, και τέλος πρόεδρε, αυτό θα ήταν δυνατότητα και με τακτική και με άτακτη αποχώρηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο και συγκεκριμένο. Να ρωτήσω, εάν έχουμε ένα ξεκάθαρο Brexit ρήξη, χωρίς διευθετήσεις για την πρόσβαση στα Βρετανικά ύδατα, πόσο θα κρατήσει για τα μεμονωμένα ευρωπαϊκά σκάφη το σύστημα αποζημιώσεων, πόσο θα αντέξει. Ευχαριστούμε. Και κύριος Φαντάλ, ευχαριστώ πρόεδρε για το σημείο 5 της σημερινής διάταξης είναι εξίσου σημαντικό με το 4. Διότι τελικά μας απασχολεί τι θα μας συμβεί στο τέλος του Οκτώβρη. Μπορεί μετά τις 31 Οκτωβρίου να υπάρχουν ε, σοβαρές εντάσεις, το βλέπουμε ήδη και από σήμερα, και επίσης μπορεί από τις 31 Οκτωβρίου εκατοντάδες αλληλευτικά σκάφη να παραμείνουν ε, πλοκαρισμένα. Οι αλληλευτικές εταιρείες θα βρεθούν πολύ στριμωγμένες. Αυτό βέβαια μπορεί να μην κρατήσει. Μπορεί μετά τον Νοέμβριο να αλλάξουν τα πράγματα. Όμως ενδεχομένως κάποιοι να κηρύξουν και πτώχευση στον τομέα τη Αλία. Η Επιτροπή μα λέει μην ανησυχείτε, έχουμε σκεφτεί όλα τα σενάρια. Όμω στην πράξη τι ακριβώ θα συμβεί. Πώ θα τι βοηθήσουμε τι εταιρείε αυτέ Θα προβλεφθούν αποζημιώσει για να αποφύγουμε μια οικονομική, ένα οικονομικό όλεθρο. Η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο τη θάλασσα είναι πολύ ωραία, Όμω ξέρετε ότι οι τέτοιε διαπραγματεύσει μπορεί να κρατήσουν μήνε και χρόνια, ενώ αυτέ οι εταιρείε μπορεί μέσα σε μερικέ μέρε να πτωχεύσουν. Θέλετε δευτερολογία. Κύριε Φαντάλ, ηλεκτρική αλεία. Έχετε αποδεκατήσει την παράκτη αλεία με την βάρβαρή σας ηλεκτροκίνητη αλεία. Οι δικές μας αποζημιώσεις τι θα γίνουν, γιατί πολύ σύντομα θα σας τη ζητήσουμε. Καλά, θέμα για άλλη συζήτηση. Μιλάμε για χρηματοδότηση. Βεβαίως υπάρχει η χρηματοδότηση από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τις εταιρείε που έχουν πρόβλημα. Το ερώτημα όμως είναι πόσα είναι αυτά τα ποσά και τι θα γίνει με αυτές τις πτωχεύσεις όταν είναι ε, πιθανό να συμβούν προσεχώς. Τώρα περνάμε σε ένα άλλο σενάριο. Μηδενική πρόσβαση στα ύδατα εκατέρωθεν. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τις διευκολύνσεις για την προπόθεση ότι μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στα Βρετανικά Η χωρί συμφωνία. Τώρα λέμε τι θα γίνει αν υπάρχει απαγόρευση πρόσβαση. Μην με παρεξηγήσετε, αλλά κανένας Ευρωπαίος ψαράς δεν χάνει αλληλευτικές ευκαιρίες λόγω αυτής της εξέλιξης. Όλοι όσοι έχουν ποσόστοση θα συνεχίσουν να την έχουν. Η διαφορά είναι ότι μεγάλος αριθμός αυτών θα πρέπει να περιοριστούν στο χώρο όπου κανονικά θα έπρεπε να ψαρεύουν τις ποσοστώσεις τους με κοινά αποθέματα κάποιες φορές ποσοστώσεις καλύπτουν ύδατα που είναι και βρετανικά και ευρωπαϊκά η διαφορά θα είναι ότι πλέον ο ψαράς δεν μπορεί να πάει στα βρετανικά ύδατα αλλά η ποσόστοση δεν θα πειραχθεί δεν ξεκινάμε συζήτηση τώρα για το πόσε ποσοστώσει θα έχει ο καθένα μεταξύ των κρατών μελών. Ούτε για του επιμέρου ψαράδε. Οι ποσοστώσει θα παραμείνουν οι ίδιε την 1η Νοεμβρίου. Ακόμα και χωρί Brexit. Χωρί συμφωνία, μάλλον, στο Brexit. Απλώ οι ψαράδε θα πρέπει να κοιτάξουν σε ποια νερά θα πηγαίνουν. Γι' αυτό πρέπει να δούμε ει βάθο την ενδεχόμενη μετατόπιση, ανάγκη μετατόπιση των ψαράδων. Βλέπουμε θα δημιουργηθούν μέχρι και hot spot. Σημεία πίεσης και έντασης όταν οι ψαράδες θα αναγκαστούν να λειτουργήσουν αλλιώς. Σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Το κάναμε από την αρχή της χρονίας αυτό. έχουμε κοιτάξει τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα αποζημίωσή του. Ρώτησε ο κ. Φαντάλε τι θα γίνει την 1η Νοεμβρίου. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή πτώχευση και να καλυφθούν από αυτό το ενδεχόμενο. Εάν υπάρξει το Brexit λοιπόν και απαγόρευση πρόσβαση στα βρετανικά ύδατα, μπορεί να υπάρξει αυτή η περίπτωση τη προσωρινή πτώχευση. Είδαμε και τι τα κράτη-μέλη σκέφτονται στι συζητήσει μα τα προηγούμενα δύο χρόνια και τα, τα περισσότερα κράτη-μέλη την κοιτάνε πολύ προσεκτικά αυτή την πιθανότητα. Χρηματοδότηση λοιπόν από το πού που μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να διευκολύνουμε την ε, ανταλλαγή πόρων μεταξύ των διαφορετικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και προετοιμαστήκαμε προσεκτικά για αυτή την κατάσταση. Ρεαλιστικά και σε, με βάση την πραγματικότητα, ναι, είναι πολύ ε, σύντομο το διάστημα, όμως 14 μήνες λέμε ότι μπορεί να χρειαστούν τα μέτρα αυτά μετά την 1η Νοεμβρίου. 9 μήνες για την προσωρινή πτώχευση. Μπορεί δηλαδή αυτό κάπως να αμβλύνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίσουμε. Τροποποιήσαμε αναλόγω το πολιτέ δημοσιονομικό στην αρχή τη χρονιά. Το είδαμε με τα κάτι μέλη για τι λεπτομέρειε των δικών του προγραμματών και σχεδίων. Αυτή είναι η δική μα η προσέγγιση. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον θα μπορέσουμε κάπω να σβήσουμε την πυρκαγιά που θα ξεσπάσει εκείνη τη στιγμή, τι πρώτε μέρε, και με την προσωρινή πτώχευση θα αποφύγουμε ίσω το απόλυτο χάος και τις εχθροπραξίε. Αυτή είναι η δική μα προσέγγιση ξεκάθαρα σε συνεργασία με τα κάτι μέλη. Είναι στατηγική τη ανάγκη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διαδικασίε ε, ολοσχερούς Διότι θα έπρεπε τότε να δούμε διορθωτικές αλλαγέ στον χώρο τη αλίας προηγουμένω. Ό,τι και να γίνει την, επο, την επαύριο του Brexit, ελπίζουμε ότι η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάρξει και θα συνεχιστεί και με αυτού κάποιο είδου συνεργασία Τότε λοιπόν δεν θα χρειαστεί να είμαστε τόσο δραστικοί στα μέτρα μας με μόνιμες πτωχεύσεις. Δεν είχε περιληφθεί στην τροποποίηση του Πουδουπού λοιπόν αυτό. Ο κύριος Γκονζάλης νομίζω ρώτησε τι γίνεται με τα σκάφη και τις σημαίες τους. Ε, τα σκάφη με βρετανική σημαία αλλά ξένοις πλειοκτησίας δεν είναι ένα θέμα που μπορούμε να το δούμε εμείς στην Αλία. Αυτό έχει να κάνει και με το μέλλον των επενδύσεων στον Ηνωμένο Βασίλειο και πόσο θα επιτρέπουν ε, τις επενδύσεις στον τομέα της Αλίας, θα τις ενθαρρύνουν. Ό,τι και να πω επ' αυτού, θα πω κάτι πολύ βλακώδες. Οπότε προτιμώ να το αποφύγω. Έγινε ερώτηση και για τις εξαγωγές. Γνωρίζουμε τι θέλουμε εμείς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολουθούμε τις προτροπές σε ένα βαθμό του Ηνωμένου Βασιλείου και γερισμένα προϊόντα βλέπουμε και δημοσιεύσεις στα ανάλογα site αλλά δεν μπορώ να σα δώσω ένα πλήρη κατάλογο των απαιτήσεων του ΕΒ τι θεωρούν εξαίρεση και τι όχι και αν είναι, πόσο είναι ικανοποιημένοι. Συζητάμε συγκεκριμένε παρεκκλήσει, αλλά όπως είπα, συνολική στρατηγική της Επιτροπής και του Μπαρνιέ, του κυρίου Μπαρνιέ, σε δημοκρατήσεις με το Brexit, είναι να μην υπάρχουν λεπτομερείς συνομιλίες ακόμα, για τις λεπτομέρειες δηλαδή. Νομίζω ότι τα απήντησα τα περισσότερα. Απάντησα πόσο καιρό, 9 μήνες, 270 τόσες μέρες. Είναι το μέγιστο για την ε, προσωρινή πτώχευση. Κυρία Μπιλμπάου, έχει απαντηθεί η ερώτησή σας. Ναι. Πρόεδρε, θα ήθελα μια απάντηση για την ερώτηση που υπέβαλα για την ε, Σκοτία. Αν αυτό αλλάζει κάτι. Ευχαριστώ. Ναι. Θα ήθελα να συζητήσω το τι θα γίνει με τη Σκωτία και το μέλλον της Σκωτίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι δουλειά μου. Ένα αυτό και δεύτερον, θα ήταν πραγματικά σκέτη κερδοσκοπία. Ε, θα ήταν σκέτη κοτολογία και εικασία να προσπαθούμε να πούμε τι θα γίνει με τη Σκωτία. Ναι, ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε. Τι έχει γίνει τρει μήνε, τρία χρόνια διαπραγματεύσεων, έξι μήνε πριν, ε, αφού το Ηνωμένο να έχει μη φύγει και πόσο καιρό μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Όλα πάλι βέβαια πλήρη ανασφάλεια και πιθανότητα τα πάντα να καταλήξουν σε απόλυτο χάο. Τίποτα δεν ξέρουμε πάλι. Πάντω, σα ευχαριστούμε που ήσασταν τόσο σαφεί, ακόμη και αν κάποιε φορέ είσαστε αρνητικό σαφεί. Σα ευχαριστούμε if we could turn to the next item. Να πάμε στο επόμενο σημείο. Τα τάκ της Βαλτικής. Ah. Mrs. Kirchner is going to give us a proper presentation. Very good. So, as you all know, uh, the, the... Ακούσουμε μια πολύ μετά όλα της παρουσίαση. Ξέρετε ότι είχαμε τις ε, συστάσεις κομισιών ε, πριν από δύο-τρεις εβδομάδες, τρία χρόνια μετά το πρώτο πολιετές ε, πλαίσιο για την Βαλτική. Θα πρέπει να γίνουν περικοπές στα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα, ΤΑΚ. Θα ακούσουμε λοιπόν το πώς μπορούμε να πετύχουμε μέχρι το 2020 τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση σύμφωνα με την κοινή αλληλευτική πολιτική, αλλά και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε την, ε, τον αλληλευτικό κλάδο. Και αν συμφιλιώνονται αυτά τα δύο μεταξύ του, κύριε Κούσνερ, έχετε το λόγο. Ε, Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περίμενα με ανυπομονησία να φορτωθεί η παρουσίασή μου για να σας την ε, προσφέρω. Μισό λεπτό να λυθεί το πρόβλημα με τις διαφάνειες. Α, ωραία. Τα καταφέραμε κάποιες γενικές παρατηρήσεις για τη Βαλτική θάλασσα. Πολύ σωστά λέτε ότι η Βαλτική είναι η περιοχή ακριβώς της Ένωσης που ήδη έχει πολιετές πρόγραμμα διαχείρισης για μια τριετία. Από την άλλη όμως ταυτόχρονα, δυστυχώς και πρέπει να το πω, είναι και η θαλάσσια λεκάνη της Ένωσης που περνάει από σοβαρές περιβαλλοντικές αλλαγές, δραματικές, πραγματική αλλαγή του μοντέλου και του παραδείγματος στην Βαλτική. Έλλειψη οξυγόνου, προβλήματα με την ε, αλμυρότητα του ε, εδάφου, των του πυθού, ε, του πυθμένα, με την ευτροφισμό και όλα αυτά βεβαίως πλήττουν τα αποθέματα. Πριν ξεκινήσω με το πρώτο είδος, την δυτική ρέγγα, να πω ότι έχουμε 10 τάκ, 10 ποσοστά μεγίστων αποθεμάτων στην Βαλτική, οπότε μας απασχολούν αυτές οι ποσοστώσεις. Από τα 10 αυτά, τα πρώτα 4 που θα σας παρουσιάσω, είναι ειδικέ περιπτώσει. Γιατί είναι ειδικέ περιπτώσει, Γιατί για τα πρώτα 4 είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι επιστήμονε θεωρούν έχουν μάλλον αλλάξει την θεώρηση του αποθέματος. Πολύ σημαντικό να το έχετε κατά νου, διότι ακριβώς για αυτό το λόγο κάποιες φορές έχουμε δραστικές μειώσεις στις προτάσεις μας. Τι εννοούμε οι επιστήμονε έχουν αλλάξει την επισκόπησή του για τα αποθέματα. Κάθε τρία χρόνια οι επιστήμονε συγκεντρώνονται και κοιτάζουν όλα τα δεδομένα που έχουν στα χέρια του για τη δυτική ρέγγα, για τον δυτικό ε, γάδο, για τον ανατολικό γάδο και ε, για την ε, ε, ρέγκα του Βοθνιακού. Και μετά Ανάλογα με την εικόνα που διαμορφώνεται, κοιτάζουμε αν οι ποσοστώσεις που προτείναμε προηγουμένω είναι σωστές και αν πρέπει κάτι να το μειώσουμε, να το αυξήσουμε. Αν πρέπει να μειώσουμε κάτι, κοιτάζουμε τι είναι αυτό. Δηλαδή, μπορεί οι επιστήμονε να προτείνουν ότι εκεί που έχουμε λιγότερα ψάρια στη θάλασσα, πρέπει να δούμε την ποσόσταση τη περσινή χρονιά. Και επειδή έχουμε πλέον επιστημονικά δεδομένα σε σχέση με την περσίνη χρονιά, βλέπουμε ότι το απόθεμα όντω ε, συρρυκνώθηκε. Ή μπορεί να πούνε ότι πριν από δύο χρόνια υπήρχε μια νέα τάξη έτους όπως το λέμε, είχε δηλαδή το απόθεμα εμπλουτιστεί με την προσχώρηση νέων ε, ε, ψαριών και τώρα εκτιμούμε διαφορετικά τη νέα τάξη έτους. Εάν οι αλείς μας πούν ότι είναι πολύ μικρότερο το απόθεμα, έχουμε πολύ λιγότερα νέα ψάρια, τότε ε, πρέπει να υπάρξει ε, αναθεώρηση προς τα κάτω. Αυτό ισχύει για τα τέσσερα πρώτα αποθέματα λοιπόν. Ξεκινάω με το πρώτο, την ε, δυτική ρέγγα. Τη ρέγγα της δυτικής βαλτικής δηλαδή. Εδώ η ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι μέχρι πέρσι Μα είπε, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τότε μα είπε το Διεθνέ Συμβούλιο για την ε, έρευνα τη θάλασσα, ότι υπάρχει ε, μείωση στο απόθεμα. Και μα είπαν κάτι δεν πάει καλά εδώ. Η βιομάζα είναι πολύ μικρότερη από ό,τι νομίζαμε. Γι' αυτό θα εκδώσουμε σύσταση μηδενικού, μηδενικής αλίευσης. Και αυτό το κάνουν κάθε φορά που βλέπουν ότι δεν υπάρχει τάκ όσο μικρό και αν είναι το ΤΑΚ, ακόμα και 5% μόνο να είναι ε, και να έχει χρησιμοποιηθεί την περασμένη χρονιά, δεν μπορούμε έστω και με αυτό να βεβαιωθούμε ότι θα πάει πάνω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο το απόθυμα του ψαριού. Οπότε, όποτε ένα απόθεμα είναι κάτω από το επίπεδο του, του, του, του κινδύνου, λένε μηδενική ποσόστοση οι επιστήμονες. Ευτυχώ που είχαμε το πρόγραμμα, γιατί με το πρόγραμμα μπορούμε να εφαρμόσουμε τις παραμέτρους του. Μπορούμε να αποφύγουμε τη μηδενική ποσόστοση, όπως έγινε με την δυτική ρέγγα ε, οι επιστήμονε για του χρόνου λένε λοιπόν ότι είναι κάτω από τα επίπεδα κινδύνου η ασφαλεία. Δεν θα επανακάμψει την ερχόμενη χρονιά. Μετά το 2022 μπορεί να επανακάμψει, το βλέπετε στη διαφάνεια. Οπότε σα συνιστούμε να μην αλλιεύσετε τίποτα. Το πρόγραμμά μα μα λέει το εξή. Ότι πρέπει να ορίσουμε τάκ ε, χαμηλού επίπεδου και ότι πρέπει να λάβουμε επιπλέον μέτρα ε, αποκατάσταση. Τι προτείνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι παρόμοιο με αυτό που είχαμε προτείνει πέρσι. Δηλαδή ένα πακέτο δύο μειώσεων ταυτόχρονων. Η πρώτη μείωση είναι μείον 42% για την ε, συνολική ποσόστοση, μείωση τη ποσόστοση λοιπόν, και μετά επιπροσθέτω μέτρο αποκατάσταση, αυτό που μα ζήτησε δηλαδή να κάνουμε ε, το Συμβούλιο, επιπλέον μείωση 29%. Θα ρωτήσετε τώρα γιατί μείον 42% και γιατί μείον 29% ε, και γιατί δεν είναι στρογγυλή αριθμή. Το μείον 42% είναι το ελάχιστο ε, που επιτρέπεται στο χαμηλότερο επίπεδο και το μείον 29% το επιλέξαμε ως αριθμό γιατί αν προσθεθούν φτάνουμε στο μείον 81%. Και στην ε, συμβουλή του ISIS λέγεται ότι το μείον 81% μπορεί και να φέρει το 2022 το ψάρι, τα αποθέματα, ε, πάνω από τα επιτρεπόμενα επίπεδα. Μέχρι το 2020 θέλουμε το απόθεμα του ψαριού να έχει φτάσει κάτω από το επίπεδο. Μείον, 71% εννοείται. Ναι, μέχρι το 2022, σωστά. Με το μείον 71% που προτείνουμε φέτος το φετινό τάκ για του χρόνου, εννοούμε ότι θέλουμε να περάσουμε το ελάχιστο επίπεδο κινδύνου. Αυτό λέει και το πρόγραμμα το πρόγραμμα λέει ότι πρέπει να αποκατασταθούν τα αποθέματα ή να αποκαθίστανται συστηματικά. Πάω στο επόμενο δύσκολο. Είναι ο ε, δυτικό γάδο, ο γάδο τη Δυτική Βαλτική. Το ίδιο και εδώ. Πριν από τρία χρόνια μα είπαν ότι υπήρχε πρόβλημα με το απόθεμα οι επιστήμονε. Είδαν τα δεδομένα και είπαν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο νομίζαμε. Ο γάδο υποφέρει. Οπότε τώρα έχουμε νέε πληροφορίε οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το 2016 είχαν μια πολύ καλή ταξία τους ε, και είχαμε πολύ, πολλά, πολλούς νέους γάδους που ήρθαν και προσχώρησαν στο απόθεμα. Φέτος όμως το ISIS e ξαναείδε προσεκτικά του συνολικούς αριθμούς και είπε ότι το μέγεθος αυτό του νέου κοπαδιού ήταν το μισό από αυτό που νομίζαμε. Οπότε έπρεπε να μειώσουμε τις προβλέψεις μας. Γι' αυτό περιμένουν σοβαρή μείωση και εμείς προτείναμε μείον 68% το ε, λιγότερο επίπεδο μέγιστου ε, βιώσιμη, μέγιστης βιώσιμης που επιτρέπεται και είναι και η τιμή που πρότεινε το ISIS στις συστάσεις του. Αυτό μας έστειλαν και είπαν ότι καλό θα ήταν να ορίσουμε το τάξη στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. 3.065 λοιπόν, τόνοι, σημαντική αριθμή γιατί αφορούν το κάνουν οι εταιρείε που εμπορεύονται τον γάδο και βλέπετε και τον αριθμό που θα επιτρέπεται για το χρόνο για τους αλείς. Η τελευταία γραμμή επίσης του, ε, της διαφάνειας λέει ότι επιτρέπονται δύο ε, σάκι με ψάρια ε, ημερησίως για τους ερασιτέχνες αλείς. Αυτό στην πράξη έχουμε υπολογίσει πόσο περίπου βγάζει πόσα ψάρια θα αλλιεύουν ετησίω οι ερασιτέχνες αλείς και αν τα προσθέσετε και τα δύο φτάνετε στο MSY, το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο αλλία. Ε, Είναι σημαντικό το Συμβούλιο να λάβει τη σωστή απόφαση αυτή, διότι το απόθεμα αυτό ε, βασίζεται μόνο σε ένα καλό χρόνο. Ε, έναν... Ε, αυτό ήταν το 2017 τότε προβλέπεται να ήρθαν πολλά νέα ψάρια, πολλοί νέοι γόνοι, αλλά μετά το 2018 ήταν μια πολύσυνη χρονιά και το 2019 δεν ξέρουμε ακόμα, θα το ξέρουμε του χρόνου. Μετά πάμε στο επόμενο, ε, τον Ανατολικό Γάδο. Αυτή είναι η πιο δύσκολη ιστορία της ε, Βαλτικής και είναι και το απόθεμα που αντιδρά Πρώτο, από όλα τα αποθέματα των ε, ψαριών στην Βαλτική, στα περιβαλλοντικά προβλήματα που έλεγα προηγουμένω. Το ψάρι αυτό, λίγε εβδομάδε πριν όταν ήμουν στην Επιτροπή σας την περασμένη φορά, λέγαμε πόσο μικρό είναι το απόθεμα. Δεν υπήρχε ε, τίποτα καλό γι' αυτό. Το σηκώτη είχε επηρεαστεί από ε, σκουλίκια. Ε, υπάρχει πρόβλημα με τον πυθμένα, έλλειψη ε, τροφής στον πυθμένα της θάλασσας. Είναι δραματική λοιπόν η κατάσταση εδώ. Τι προτείνουμε για το χρόνο. Προτείνουμε να κλείσουμε όλα τα τάκ για τον Ανατολικό Γάδο. Και το ISIS λέει μηδενικά αλλιεύματα. Μην ψαρεύετε γάδο τα μηδενικά λεύματα για τον γάδο τη Ανατολική Βαλτική. Τι θα γινόταν το προτείναμε ακριβώ έτσι. Θα έπρεπε να κλείσουμε κι άλλα αλλιεύματα. Να τα αποκλείσουμε, δηλαδή τη χωματίδα, την πελαγική Αλία, διότι όλα αυτά έχουν και λίγα παραλιεύματα ανατολικού γάδου. Ε, αντί λοιπόν να τα κλείσουμε και όλα τα άλλα μαζί, είπαμε κλείνουμε τη στοχευμένη αλία γάδου και επιτρέπουμε ένα ελάχιστο επίπεδο 2.000 τόνων, ποσό που όταν το υπολογίσαμε είναι τα παραλιεύματα που δεν μπορούν να αποφευθούν μαζί με, την αλλιεύση άλλων ειδών, δηλαδή τα άλλα μπορούν να συνεχίσουν να είναι οικονομικά βιώσιμα, να συνεχιστούν οι ελεκτικές δραστηριότητε, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουμε τουλάχιστον το γάδο. Και λέμε δεν, το, δεν μπορείτε να το στοχεύετε. Κάτω τα χέρια από το γάδο. Επίσης, ένα επιπλέον μέτρο είναι κλείσιμο για την περίοδο οτοκίας. Αυτό το προτείνουμε από τον Μάιο ως τον Αύγουστο για όλα τα σκάφη σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή. Η ιδέα είναι να επιτρέψουμε σε αυτή την περιοχή που ξέρουμε ότι υπάρχει οτοκία να είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε όχληση. Ελπίζουμε ότι με την πάραδο των ετών, όχι για ένα χρόνο, το προτείνουμε για τα επόμενα χρόνια που ακολουθούν. Ελπίζουμε ότι τα επόμενα λοιπόν χρόνια το μέτρο αυτό, αυτή η πάυση της αλίας, αυτή η αλληλευτική πάυση θα επιτρέψει να αποκατασταθεί το απόθεμα. Και λέμε και στους ερασιτέχνες αλληλείς, αυτούς που ψαρεύουν με καλάμι, δεν μπορείτε στις περιοχές 25 και 26, όπως τα βλέπετε στην τελευταία γραμμή, να ψαρεύετε άλλο με καλάμι. Εδώ δεν μπορούμε να τους εξηγήσουμε μην ψαρεύετε με, καλά, με τον γάδο ειδικό, μην ψαρεύετε σε αυτές τις περιοχές τους λέμε. Και αυτό έχει βεβαίω και αντίκτυπο στα, λιεύματα, στα αποθέματα των ψαριών στη Βαλτική. Πάμε στο επόμενο τώρα, τη ρέγγα του Βοθνιακού. Εδώ έχουμε μια παρόμοια κατάσταση. Απειλείται η ρέγγα. Αλλά όπω και για τα προηγούμενα δύο, ε, το Συμβούλιο Έσχη άλλαξε άποψη. Μα είπαν κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώ τι ακόμα. Λένε πάντω ότι κάτι σε σχέση με τα δεδομένα δεν πάει καλά και λένε ελπίζουμε να το βρούμε ακριβώς του χρόνου, να το εντοπίσουμε. Τώρα είναι θέμα βιομάζας, είναι θέμα της πίεσης από την αλία. Θα το ξέρουμε σίγουρα του χρόνου. Όμως, ακριβώς επειδή έχει ενδιασμού στο ISIS, τι έκανε. Άλλαξε και την ποιότητα της Συμβουλής. Μέχρι τώρα είχαμε μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο αλίευσης. Αυτό που είχαμε από το 2019. Επειδή όμως τώρα έχουμε συμβουλή πρόληψης, πρέπει να μειώσουμε και την ποσόστοση για το 2019 ήδη. Οπότε πάμε στη συζήτηση που είχαμε και πέρσι, μάλλον πριν από λίγες εβδομάδες, όταν κάποιοι από εσά λέγατε γιατί δεν επιτυγχάνουμε, προσπαθούμε να έχουμε μέγιστο απόθεμα για τα 200 είδη που πραγματευόμαστε, γιατί το κάνουμε μόνο για ένα, το κάνουμε εκεί που έχουμε συμβουλή μέγιστο επίπεδο αλλίευση. Εδώ είναι η απόδειξη. Το ISIS μα λέει δεν μπορούμε να σα πούμε ποιο θα ήταν το MSY, μπορούμε μόνο να σα δώσουμε μια συμβουλή πρόληψη. Γι' αυτό λοιπόν βγαίνει από τον κατάλογο MSY. Δυστυχώ. Γιατί εδώ θα μα συνέφερε πολύ να έχουμε συγκεκριμένη εικόνα. Οπότε αναγκαστικά προτείναμε μείωση. Πάμε στο επόμενο. Η κεντρική ρέγγα και η σαρδελόρεγγα. Εδώ έχουμε διαφορετικά είδη αποθεμάτων. Τα πρώτα σας τα έχω ήδη παρουσιάσει και είπα ότι έχει αλλάξει εδώ η εικόνα μας για το τι συμβαίνει. Τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Προτείνουμε και πάλι μειώσεις, το βλέπετε, η κεντρική ρέγγα είναι μείον 10%, σερδελό ρέγγα μείον 25% και όχι γιατί υπάρχει αλλαγή στο τι συμβαίνει με τα ψάρια στην πραγματικότητα, το βλέπετε με πράσινο κάτω. Ε, μόνο ένα καλό ε, έτος τάξης είχαν τα ε, ψάρια αυτά Οπότε τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Να αφήσουν περαιτέρω χρόνο στα ψάρια αυτά της καλής χρονιάς, ώστε να ανανεωθούν οι γόνοι και τα αποθέματα. Θέλουμε να αφήσουμε δηλαδή λίγο χρόνο και να δούμε τι συμβολή θα δώσει το ISIS του χρόνου. Ε, εδώ οι μειώσει δεν είναι επειδή καταραίει το απόθεμα, περιορίζεται και συρρυκνώνεται, αλλά γιατί έχουμε μόνο ένα καλό έτος. Τα επόμενα έτη μετά από την καλή αυτή χρονιά δεν ήταν τόσο καλά και έτσι προκύπτουν οι μαθηματικοί υπολογισμοί του ΆΕΣΑ. Και πάμε στο επόμενο, τη χωματίδα, η πλατέσα. Έχουμε μια ποσόστοση, αλλά αυτή έχει διαμορφωθεί από δύο διπλές συμβουλές. Η μία είναι το μέγιστο επίπεδο αλίευσης, επιτρεπόμενο επίπεδο αλίευση. Και το άλλο μικρότερο κομμάτι τη ποσόστοση είναι ε, συμβουλή προληπτική. Πρέπει να συνδυάσουμε και τα δύο για να καταλήξουμε σε μία ποσόστοση, αυτή που βλέπετε, και πάμε στο μείον 32%. Εάν το Συμβούλιο ακολουθήσει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε η μείωση θα φτάσει το μείον 32% και θα συνεχίσει να καταγράφεται και ω είδο MSY, με μέγιστο επίπεδο αλίευση. Μετά πάμε στους δύο σολομούς που έχουμε στην Βαλτική. Ο ένας είναι ευτυχώ MSY, μέγιστο επίπεδο αλίευσης, ο άλλος όμως του κόλπου της Φινλανδίας έχει και πάλι ε, προληπτική ε, αποτίμηση. Ελπίζουμε να πάρουμε μέγιστο επίπεδο από θέματο MSY του χρόνου. Ε, είναι πάντως καλό επίπεδο, είναι καλό είδος για MSY αλλά εδώ μπορούμε να προτείνουμε μετακύληση. Ε, εδώ λοιπόν η αλληλευτική πίεση είναι κάπως υψηλή. Προτείνουμε μείον 5% και είναι σημαντικό για το Συμβούλιο να δούμε αν θα μας ακολουθήσει ή αν θα προτιμήσει μετακύληση. Μετά για το Σολομό του κόλπου της Φιλανδίας, το ίδιο ισχύει και εδώ. Ακολουθούμε μία ε, επιφυλακτική προσέγγιση. Είχαμε μειώσει το, το, το τάκα από πέρσι εδώ έχουμε μόνο μια καλή ιστορία, μια θετική με αύξηση στην ποσόστοση για την ε, Βαλτική και αυτή είναι η ρέγγα της Ρήγας. Είναι το μόνο είδος με αύξηση. Είναι σε καλή κατάσταση ε, και με, ακόμα και με, αν με αύξηση 11% θα παραμείνει ένα ψάρι με μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ε, πρόεδρε, για το που έχουμε φτάσει λοιπόν με, τα μέγιστα, ε, με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για το 2020 βλέπετε ότι έχουμε θεωρήσει έξι από τα είδη να είναι σωστά σε σχέση με τις απαιτήσεις της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και έχουμε και κάποια τάκ για τα οποία έχουμε μόνο μια προληπτική προσέγγιση, διότι δεν μπορούμε και γι' αυτό δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα το δείτε στη δεύτερη ε, γραμμή, είναι η ρέγγα του Βοθνιακού και ο Σολομός του κόλπου της Φιλανδίας. Εκεί περιμένουμε να δούμε τι στοιχεία θα συγκεντρώσουμε του χρόνου και τα τελευταία, δύο, τα τελευταία δύο είναι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις. Η ρέγγα του, της Δυτικής Βαλτικής και ο Γάδος εδώ δεν έχουμε εκφορτώσεις και δεν έχουμε καταγράψει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ακόμη και αν το Συμβούλιο αποφασίσει μηδενική ποσόστοση για του χρόνου, κάτι δεν πάει καλά σημαίνει αυτό, δεν μπορούμε να τα βάλουμε στον κατάλογο του MSY. Έξι από τα οκτώ λοιπόν Αυτά που θα έπρεπε να είναι στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση περιλαμβάνονται, τα άλλα θα περιμένουμε το 2020. Θα έλεγα να πάψω εδώ και μετά να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος τα προηγούμενα χρόνια είχε υποστεί κριτικές που δεν ακολούθησε τις ε, επιστημονικές συμβουλές. Άρα πολύ χαιρόμαστε που εσείς τις ακολουθείτε. Ο αντίκτυπος για τις θέσεις εργασίας ε, στην Παλτική είναι σημαντικός. Σοβαρός θα έλεγα. Είχαμε νέες επιστημονικές αξιολογήσεις ε, που έδειξαν ότι το απόθεμα δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση όσο αυτό που νομίζαμε. Το σκουμπρί του Βορειοατλαντικού π.χ. φαίνεται ότι είναι περισσότερο από ό,τι έδειχναν οι επιστημονικές ενδείξεις. Και με οποιοδήποτε σφάλμα υπάρχουν απώλειες θέσεων απασχόλησης. Δεν περιμένω απάντηση από εσά, απλώς ε, όταν μιλούμε για τόσο συνολική περικοπή της ε, συνολικής βιομάσας, δεν είναι, κάτι, δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς ε, μετά από ένα πολιετές σχέδιο διαχείρισης και την εφαρμογή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως μία ερώτηση, πολλά ακούσαμε, έχουμε μία δύσκολη πραγματική κατάσταση στην Βαλτική και δεν είναι μόνο η υπεραλίευση, είναι λίμανση, ε, ρήπη, ε, ε, κλιματική αλλαγή κτλ. Πίσω από τα μεγέθη αυτά πάντως υπάρχουν υπάρχει και η απειλή για τις ε, θέσεις απασχόλησης. Η Επιτροπή νομίζω ότι είχε στη θέση της 1,5 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ ώστε να αναπτύξει ένα κέντρο παραγωγής υψηλού επίπεδου και ξαφνικά απειλείται με κλείσιμο. Εάν ε, εφαρμοστεί το κείμενο αυτό ε, απειλούνται με εξαφάνιση οι μικροί στόλοι, τα μικρά σκάφη και όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά και για τη Δυτική Ρέγγα και για το Δυτικό Γάδο. Στη περιοχή 24, αν διερθεί στα δύο, θα μπορούσε να εξετάσει κανεί δυνατότητε ε, λίγο υψηλότερης αλίευση, ιδιαίτερα του Δυτικού Γάδου. Ιδιαίτερα για τη Δυτική Ρέγγα είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα για τις παράκτιες ζώνες που ενέχονται είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πρέπει βεβαίως να εξετάζουμε και να λαμβάνουμε σημαντικά υπόψη τι λένε οι επιστήμονες, αλλά όταν σφάλουν, όπως είπε και ο πρόεδρος, τότε είναι ανεπανόρθωτη η βλάβη. Πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη μας τι σημαίνουν όλα αυτά για τις παράκτιες κοινότητες τις αλλιευτικές. Ίσως οι μειώσεις να μην είναι τόσο σημαντικές όσο αυτές που μας παρουσιάσετε. Ε, η κυρία ε, Κούσνα θα πρέπει να, να αναφερθεί και στο τι θα συνέβαινε αν δεν γινόντουσαν δεκτές οι συστάσεις της. Ίσως ε, πρέπει να είμαστε σκληροί ώστε να είμαστε ευγενικοί, αλλά ενέχονται και άνθρωποι και οι δουλειές τους όπως ακούσατε. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την απειρά αλλά και το τι αποφάσεις θα λάβουμε και ελπίζουμε από την Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει σωστά και να δούμε πού είναι το πραγματικό πρόβλημα με την αλία στη Βαλτική. Το θέμα είναι τι ρεαλιστική προσέγγιση θα ακολουθήσουμε όπως θέλει να το πει κανεί. Από τη στιγμή που έχουν υποβληθεί οι προτάσεις αυτές, εγώ βρίσκω ότι η κατάσταση είναι ακόμη πιο κρίσιμη. Και το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή για να βοηθήσει τον κόσμο εκεί πέρα θα κάνουμε για το μέλλον τους. Είναι δυνατόν να υποστηρίξουμε την αλία με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έχουμε ήδη ακούσει τις υπελιγμούς για το πολιτής δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά θέλουμε να δούμε και βραχυπρόθεσμα τι μπορούμε να κάνουμε. Για αυτούς που δεν έχουν καμία πρόσβαση στην αγορά. Έχει σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετικά τι μπορεί να αλλάξει ώστε να βοηθήσουμε κόσμο που μπορεί να έχει πρόβλημα με τη δουλειά του και δεν μπορεί να βοηθηθεί από τα κρατη Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τον ε, τουρισμό που μπορεί να πληγεί. Στις, ε, τον τουρισμό που έχει σχέση με λιμάνια και αλεία. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πολλές εταιρείες θα πληγούν όχι μόνο στη Γερμανία ή την Δανία, αλλά γενικώ στις χώρες που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Λέμε για επιστημονικές συμβουλές και γνώσεις, αλλά στη Γερμανία πολλοί ισχυρίζονται ότι οι συμβουλές για μείωση δεν είναι, οι μειώσεις που προτείνονται δεν είναι απαραίτητες. Και ο παράγοντας του τουρισμού βλέπουμε ότι τα επίπεδα μείωση που προτείνονται πλήττουν πολλέ φορέ τον τουρισμό. Πώ θα, πώς θα φροντίσουμε να παραμείνει ελκυστικό ο τουρισμό εκεί, και είναι κρίμα που δεν το έχουμε δει ω τώρα. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκεφτεί κάποια είδου μεταβατική λύση για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Σουάλβαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι ανησυχητικά ε, τα στοιχεία, τα επιστημονικά και ο πολυεπίπεδος αντίκτυπος ε, που έχει η αλίευση στην βιομάζα Μία ερώτηση είχα προς την εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν για την ανάκτηση, την ανοικοδόμηση του αποθέματος μέχρι το 2022. Ο, ο κοινό στόχος της ΚΑΠ είναι να αλλιεύουμε εντός του MSY, δηλαδή εντός της ε, μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Πώς θα επιτύχουμε την μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Διότι αυτό είναι ο στόχος που έχει προσυπογράψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, κοιτώντα τα αποδεικτικά στοιχεία, τις ενδείξεις, υπάρχει πολύ σημαντικό πρόβλημα στο μέλλον και για τη βιομάζα και γενικώ για τους αλληλείς. Η Κομισιόν λοιπόν τι σκοπεύει να κάνει προκειμένου να αυξήσει τα επέδα της βιομάζας. στην συνάντηση του Συμβουλίου τον Οκτώβριο θα υπάρξουν κάποιες ε, μνήες στις ε, μετακινήσεις ή τις εγκαταλείψεις των ε, αλληλευτικών περιοχών διότι και αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο επί των αποθεμάτων της δυτικής Βαλτικής. Σε γενικές γραμμές λοιπόν τι σχεδιάζει να κάνει η Κομισιόν προς τον μακροπρόθεσμο στόχο της ε, μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Αυτά που μας δείχνουν τα επιστημονικά στοιχεία είναι μια τεράστια κρίση. Η Κομισιόν εδώ εξετάζει το ελάχιστο δυνατό επίπεδο, αλλά αυτό δεν επαρκεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στοχεύει στο MSY και όχι σε κάτι χαμηλότερο από αυτό. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και τι γίνεται όμως για την, ε, με την ε, ρέγγα της Ρήγας και άλλα είδη της Βαλτικής που υπήρξαν επιτυχή παραδείγματα. Γιατί είναι τόσο διαφορετική η κατάσταση με τα ε, είδη αυτά. Άλλες ερωτήσεις έχουμε, λέει ο πρόεδρος. Η ρέγγα της Ρήγας λοιπόν, μήπως είναι αυτή η χρυσή λύση και το MSY αυτό που υπόθηκε δεν είναι μόνο η αλής. Η κυρία Κούσνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπάθησω να απαντήσω μία προς μία τις ερωτήσεις. Καταρχάς, στον Τι το εργοστάσιο, το λευτικό, ήρθαμε σε επαφή μαζί τους. Υπάρχουν μεγάλες ε, μειώσεις ε, που προτείνονται για τη Δυτική Ρέγκα την Κομισιόν. Μεγάλη ιστορία γιατί το ΤΑΚ αυτό το ε, μειώσαμε κατά το ίμιση και πέρυσι. Αν ξέρουμε ότι από θέματα δεν θα περάσουν τα όρια, το όριο το 2021, που μπορεί ήδη να περιμένει ότι το ISIS και το χρόνο θα πεινεί δεν, δηλαδή ξέρουμε ήδη ότι θα πρέπει να προτείνουμε μεγάλη μείωση και για το χρόνο. Δυστυχώ έτσι ε, δουλεύουν αυτά τα σχέδια. Όταν είναι κάτω του επικίνδυνου επίπεδου το απόθεμα, που δεν θέλουμε να φτάσει δηλαδή, για να μην καταρρεύσει και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Όσο λοιπόν είναι κάτω σε αυτό το επικίνδυνο επίπεδο, πάντοτε θα είναι αυστηρές οι προτάσεις. Όχι μηδέν, αλλά πάρα πολύ μεγάλες περικοπές θα προτείνονται. Νομίζουμε ότι γενικά πάντα είναι καλό τα ε, στάσια μεταποίησης να μην βασίζονται μόνο σε ένα απόθεμα, αλλά να έχουν και κάποιες αναλλακτικέ. Πρέπει να δούμε αν το συγκεκριμένο κλάδο θα μπορούσε να παίρνει πρώτε σύλλε από τη Βόρεια Θάλασσα, από άλλα αποθέματα που τα πηγαίνουν καλύτερα. Υπάρχουν στη Βόρεια Θάλασσα άλλε ρέγγε που τα πάνε πολύ καλύτερα σε σχέση με τη Δυτική. Επίσης, είπατε την περιοχή 22 γιατί να μην τη διαιρέσουμε σε δύο περιοχές για να επιτρέπουμε περισσότερη λίγο στο δυτικό τμήμα και λιγότερη στο ανατολικό. Με τα χαράς να το κάνουμε αυτό. Χρειαζόμαστε όμως επιστημονικές συμβουλές, κάτι που δεν έχουμε προς το παρόν. Ξέρουμε ότι το Συμβούλιο ε, των, ε, της Εξέρμης Θαλασσών το βλέπει και το, το 24 θα δούμε κάτι. Ίσως και από του χρόνου να μπορούν να μας πούνε. Πού είναι η διαχωριστική γραμμή γιατί εμείς δεν ξέρουμε πού να τη χαράξουμε αν κάνουμε αυτή την υποδιέρεση. Ενδιαφέρουσα ιδέα. Δεν και μακάρι να έχουμε την επιβεβαίωση του χρόνου από τους επιστήμονες, αλλά όπως καταλαβαίνετε θέλουν χρόνο αυτά τα πράγματα. Να έρθω σε κάτι άλλο. Ο κύριος να αντιδράμε μόνο με αλληλευτικά μετά δεν αρκεί, λέτε, και το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να το δουν ολιστικά το θέμα. Ήδη από την αρχή είπα ότι έχουμε μεγάλα προβλήματα με τα ε, φωσφορούχα, τα οποία, ε, τα ζωτούχα, τα οποία ε, έρχονται και εισδύουν μέσα στο έδαφος και από τη Βόρεια Θάλασσα. Δεν υπάρχει ανταλλαγή υδάτων μεταξύ Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας και τα κράτη-μέλη πρέπει να φροντίσουν η περιβαλλοντική νομοθετία όπως αυτή για τα ζωτούχα να εφαρμόζεται. Υπάρχουν στο πλαίσιο του τρέχοντος πολιετούς να υπάρξει βοήθεια μέχρι να στο επόμενο ε, πολιετές αυτή τη στιγμή γίνει υποδιαπραγμάτευση. Και ξέρετε ότι σε αυτό το νέο πολιετές η Κομισιόν προτείνει και της δυνατότητα μόνιμης ε, από ξύλωσης ή κατάργησης. Προσωρινή πάυση δραστηριοτήτων επιτρέπεται μέχρι στιγμής. Κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν τι άλλες ποσοστώσεις είναι διαθέσιμες να δούμε. Δηλαδή μπορούμε να επαναπροσανατολίσουμε στόλο για άλλες δυνατότητες αλλίευσης, για άλλα είδη που μπορούν να αλλιεύονται με ποσοστώσεις Υπάρχουν στην Παλτική όμως ε, και άλλα είδη όπως ε, το καλκάνι και άλλα. Είναι θέμα πολύ σημαντικό. Και προκαλεί έντονα συναισθήματα. Πριν από δύο χρόνια είχαμε δει τι ε, μπορεί να γίνει με τα διάφορα είδη τα οποία ε, αλλιεύονται όταν ο έμπορος μπορεί να τα εκφορτώνει γιατί άλλοι πρέπει να τα απορρίπτουν. Το ISIS ε, έχει βάλει κάποιες ε, γραμμές. Ε, είχε τεθεί θέμα με το λαβράτι κατά το παρελθόν. Λοιπόν, εδώ έχουμε 68% για τον, 60 κάτι για τον έμπορο, τον, επί, τον αλία που το έχει ως εμπορική οικονομική δραστηριότητα το ψάρεμα. Και για τους άλλους είναι 2-2 κάτι back limit για τους εραστέχνες και το έχουμε κατεβάσει στα 2% το όριο αυτό. Το Συμβούλιο το ISIS είναι αυτό που θα ορίσει τα όρια. Αλλά αν αρχίσουμε να παίζουμε τα νούμερα, αν ανεβάσουμε το back limit, τότε έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο από αυτό το οποίο λαμβάνουν υπόψη την εμπορική αλία. Οπότε θα πρέπει εκεί να πέσουν οι αριθμοί, τα ποσοστά. Δεν μπορούμε να τα αυξάνουμε όλα. Θα είναι δύσκολο. Και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη. Υπάρχουν μισθωμένα ε, σκάφη, ναυλωμένα σκάφη που φέρνουν προσθέμενη αξία. Αλλά και από άλλες δυνατότητες μπορεί να έχουμε ε, κέρδος, όπως πρακτικές αποδέσμευσης ε, αλλιευμάτων τι θα πει να έχουμε αυτό το μπακλιντό, ποιος ε, ε, αεραστέχνης αλίας ε, ψαρεύει μπορεί να κρατήσει 7 ψάρια και να τα πάει σπίτι του. Τι τα κάνεις βέβαια τα 7 ψάρια, είναι μια ερώτηση. Δεν μπορείς να τα πουλήσεις, μπορείς να τα κρατήσεις για ίδια κατανάλωση. Άρα τελικά είναι ένα χόμπι, γίνεται για αναψυχή. Άρα μπορεί κανείς να μπορέσει να ασκήσει αυτό το χόμπι απλά με αυτό το μικρότερο όριο. Αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν. Το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει απόφαση όμως τελικά. Υπήρχε μια ερώτηση τώρα για το πώς ε, ενημερώνται, εμπλέκονται οι εμπλεκόμενοι στις προτάσεις Κομισιόν. Τους έχουμε ζητήσει να, από τον Ιούνιο να μας στείλουν τις απόψεις τους. Τότε κάναμε το λεγόμενο policy statement. Είναι ένα έγγραφο που ε, δημοσιεύουμε κάθε χρόνο αφού έχουμε μιλήσει με τα γνωμοδοτικά συμβούλια, τους εμπλεκομένους φορείς, τα κράτη-μέλη και λέμε σε όλους στείλτε μας απόψε σας. Δείτε τις επιστημονικές συμβουλές, πείτε μας τι προτείνετε για του χρόνου. Και τους συναντήσαμε τους εμπλεκόμενους ε, και στις αρχές Σεπτεμβρίου όπου είδαμε την πρόταση μαζί τους ε, στο Ελσίνκι, στο πλαίσιο της συνεδρίασης των, ε, του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική. Το επόμενο, πώς θα πετύχουμε τη μέχρι με απόδοση που θέλει το Κοινοβούλιο, μια διευκρίνηση ίσως. Μάλλον κάποια παρανόηση υπήρξε εδώ. Γιατί μιλήσατε ότι έχουμε επιλέξει τη μέχρι στιγμή που έχει κάτι κατώτερο ω επίπεδο. Όχι, ακούστε. Εμείς έχουμε κάποιες περιοχές τιμών, έχουμε μια χαμηλότερη βιώσιμη ανάπτυξη και έχουμε και την ε, μέγιστη βιώσιμη ανάπτυξη. Και έπειτα έχουμε την ανώτερη περιοχή τιμών. Το σχέδιο τι λέει, αν έχει ένα πρόβλημα με κάποιο απόθεμα, το βάζει και στην κατώτερη περιοχή τιμών. Αυτό το συμφωνήσατε μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών. Είναι νόμιμη υποχρέωση που έχουμε. Πρέπει να κάνουμε μια πρόταση στο πλαίσιο της κάτω τιμής, κάτω περιοχής τιμών. Αυτή είναι περιοχή όμως, όπως είπα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια περιθώρια λιγμών. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας όμως ότι πολλά από θέματα βασίζονται μόνο σε μια καλή χρονιά. Αν το Συμβούλιο δεν πάρει του χρόνου την επόμενη την σωστή απόφαση, υπάρχουν επιπτώσεις για τα προσεχή έτη. Τα έχουμε δει. Πολύ δύσκολε καταστάσει έχουμε ζήσει στον Ατλαντικό. Βόρεια... That stock was threatened by collapse only 10 years ago. Ένα είδος ε, ε, γάδου, ε, Northern Hake, καταφέρουμε να καταστήσουμε το απόθεμα με τη συνεργασία όλων. Αν αυτό μπορέσαμε να το κάνουμε με ένα είδος, μπορούμε να το κάνουμε και με άλλα. But to rebuild the stocks, the decision... Η απόφαση λαμβάνεται τον Οκτώβριο ε, από το Συμβουλίο και πρέπει να είναι η σωστή. Μπορεί να είναι δύσκολη, να πονάει κάποιος, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται. Οι σωστές αποφάσεις των προηγούμενων ετών οδήγησαν στην επιτυχία που έχουμε πολλά αποθέματα τώρα. Και γιατί είναι επιτυχία η ρέγγα της Ρήγας και όχι ε, άλλες Ωραία ερώτηση. Αν είχα έρθει πριν ένα χρόνο, θα είχατε ακούσει προτάσεις για αύξηση, γιατί μπορέσαμε να αυξήσουμε για πολλά είδη πέρυσι. Γιατί φέτος όμως έχουμε μείωση τόσο πολύ. Νομίζουμε ότι είναι ατυχές το γεγονός και οφείλεται σε μία ε, συγκυρία. Υπολογίζεται πόσα ψάρια υπάρχουν, πόσα νέα ψάρια προστέθηκαν με τη νέα τάξη και ποιες είναι οι αλληλευτικές πιέσεις. Διότι κάποια ψάρια έχουν μια καλή χρονιά μόνο και πρέπει τώρα να φροντίσουμε όταν προτείνουμε μείωση να οδηγήσει σε βιώσιμη αλεία. Όταν έχουμε μείον 25 δεν σημαίνει ότι απειλείται το απόθυμα δεν είναι βιώσιμο. Το είδος είναι. Αλλά για να μείνει και του χρόνου πρέπει να μειωθεί το ποσοστό. Και ελπίζω του χρόνου να έρθω να σας τα πω πολύ πιο ρόδινα τα πράγματα. Και να έχουμε και για τη βαλτική αύξηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Χέρπστ. Ναι. Με τον υπολογισμό που κάνετε για τον back limit, και αν κατάλαβα καλά, υποθέτεται ότι ο ε, τουρισμός αλίας και η εμπορική αυτή αλία είναι το ίδιο και το αυτό. Μα δεν είναι έτσι, με αυτό το ένα προ ένα και μια ρητορική ερώτηση αν κατά το παρελθόν ε, υπήρχε η ίδια αντιμετώπιση των δύο αυτών κλάδων ε, φυσικά αν αυξηθούν τα ποσοστά εραστικής αλίας ε, δεν μπορούν οι υπολογισμοί αυτοί να συνεχίσουν να ευσταθούν. Υπάρχει πρόσθετα, υπάρχουν πρόσθετα αλλιεύματα. Αν έχουμε 7 back limit ε, και πρέπει να παραμείνει χαμηλότερο το βιώσιμη, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό το ένα προς ένα, η αντιμετώπιση σαν να είναι δύο ίδια πράγματα, δεν είναι σωστή να επανέλθω σε αυτό το αληφτικό εργαστήριο, λέει ο Να επανέλθω λοιπόν σε αυτό το ε, ε, κέντρο παραγωγής ε, το καινούργιο και τις θέσεις απασχόλησης, τις απώλειες θέσεων που θα μπορούσαμε να έχουμε εκεί. Το ετήσιο απόθεμα ήταν να αυξηθεί σε 125 από 100.000 τόνους. Αυτό δεν το κατανοώ απολύτως στην παρουσίασή σας, αλλά ότι δεν υπάρχει βιολογικός βιολογική ε, αιτίαση να μειώσουμε την ποσόστοση. Ναι, Πρόεδρε, να σας πω. Μας ζήτησαν, μας ρώτησαν γιατί δεν προτείνουμε απλά μείον 25%. Το σχέδιο έχει οικοδομηθεί, οικοδομηθεί με, με έναν τρόπο που ίσως οι ενδιαφερόμενοι φορείς δεν το κατανοούν εύκολα. Το μείον 25% εδώ δεν γίνεται διότι απειλείται το απόθεμα. Είναι κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα. Όταν ένα απόθεμα είναι κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα, πρέπει κανείς να προτείνει κάτι μεταξύ του MSY point και MSY lower, το οποίο δεν είναι μείον 25%, είναι ένα τελείως διαφορετικό μέγεθος. Προσπαθήσαμε στον Γκίλι, λέει, να του το εξηγήσουμε αυτόν, σε αυτό το νέο εργοστάσιο που έχουν φτιάξει. Γιατί πριν από τρία χρόνια είχε εγκριθεί το σχέδιο και πρέπει να εφαρμοστεί. Υπάρχει ένα μικρό περιθώριο, αλλά καθότι αυτό το απόθεμα μόνο το, μετά το 22 θα ανεβεί από το επίπεδο του MSY Point, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ποια ήταν το τάκ που είχε συμφωνηθεί το 2020 το οποίο θα διοχετευτεί στον υπολογισμό για τα επόμενα χρόνια. Είναι δύσκολη η κατάσταση, μακάρι να είχα καλύτερη δυνατότητα απάντησης να σας δώσω, αλλά δεν έχω. Αυτές είναι οι επιστημονικές συστάσεις που έχουμε λάβει και που θα εφαρμόσουμε και αυτή, εν πάση είναι η πρόταση Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. φορέ φορές έχουμε ζητήσει να ακολουθείτε τι υποστημονικέ συμβουλέ. άρα δεν μπορούμε να σε επικρίνουμε που το κάνετε. Ε, θα θέλαμε να μα ενημερώσετε για τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και πώ θα πάνε στου επόμενου μήνε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά ακόμα, λέει ο πρόεδρο και ένα ακόμα σημείο που είναι το 7. Οι συμφωνίες με το ΣΑΟΤΟΜΕ και και Πρίνσιπε η Κομισιόν έχει λόγο και πάλι. Καλό σας απόγευμα, λέει ο Μιλήτρια. Μια και είναι 12 και 20. Είμαι η νέα επικεφαλής ε, για τις αλληλευτικέ συμφωνίες και διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρε. Ήρθα εδώ να σας παρουσιάσω το νέο πρωτόκολλο και η νέα συμφωνία που διαπραγματευθήκαμε με το ΣΑΤΟΜΕ. Ολοκληρώσαμε τον Απρίλιο και τώρα συζητείται στο Συμβούλιο η πρόταση. Επί τη βάση εντολής που είχαμε λάβει ήδη από το 2017, το παρόν πρωτόκολλο εξέπνευσε το Μάιο του 2018, δηλαδή περί τον ένα χρόνο δεν είχαμε ακόμα ε, δραστηριότητα αλλιευτική. Μιλούμε για τον τόνο και μόνο και ως ε, μέρος του δικτύου Ατλαντικού και Αφρικανικών ακτών, παρακτήρων υδάτων. Μιλούμε για νέες αλληλευτικές δραστηριότητες όπως και το προηγούμενο πρωτόκολλο. 28 παραγαδιάρδικα και 6 γρηγροί. Με συνολική, συνολικό μέγεθος αναφοράς 8.000 τόνους. Πήγαμε σε 440.000 ευρώ το χρόνο ετήσια ε, τομεακή βοήθεια, εκτός από τους 8.000 τόνους. Επομένως, αυτό έχει συνολικό αντίκτυπο 400.000 ευρώ για τον ευρωπαϊκό περιοπολογισμό. Η διάρκεια του πρωτοκόλλου προηγουμένως αναδια πραγματεύεται κάθε τέσσερα έτη, τώρα θα είναι πέντε έτη που είναι καλό και για την τρίτη χώρα και δημοσιονομικά ως προς σταθερότητα αλλά και για το στόλο της και τα σκάφη της ε, θα γνωρίζουν πόσο και πού μπορούν να αλλιεύσουν. Η συμφωνία λοιπόν αυτή τη στιγμή συζητείται όπως σας έλεγα στο Συμβούλιο. Προβλέπεται 16 Οκτωβρίου να πάει στην Κορεπέρ. Η υπογραφή προβλέπεται επίσης εντός του Οκτωβρίου η συμφωνία προβλέπεται μετά την υπογραφή και από το Κοινοβούλιο να ισχύσει. Μπορώ να σας πω περισσότερε λεπτομέρειε βεβαίω για τη συμφωνία, αλλά είμαι στη διάθεσή σα αν έχετε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος, η κυρία Μπιλμπά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα απλώς ε, να πω ότι με αυτήν την νέα ανανέωση της συμφωνίας ε, που ελπίζουμε ότι θα εγκρίνει το Συμβούλιο, να σημειώσω ότι το προηγούμενο πρωτόκολλο είχε εφαρμοστεί με αρκετά μεγάλη επιτυχία και για τα δύο μέρη και για τους αλληλείς ε, των φινοειδών. Εμείς έχουμε σημαντική τέτοια ποσόστοση σκαφών και υπό την έννοια τη βιωσιμότητα είναι σημαντική η συμφωνία. Ήθελα λοιπόν να σημειώσω καταρχάς το στόχο της βιωσίμου διακυβέρνηση των υδάτων αυτών και οικονομικής βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής που είναι σημαντική και για τον δικό μας τομέα τον ελευτικό αλλά και για τον δικό τους και τη ευρύτερη περιοχή Και μόνο όλα τα μέτρα συνεργασία για την ανάπτυξη του αλλιευτικού τομέα στην περιοχή αυτή είναι πολύ σημαντική. Σε κάποια άλλα πρωτόκολλα είχαμε συμπεριλάβει και μία μνήα στην γυναικεία συμμετοχή στον τομέα. Δεν ξέρω αν και εδώ είχαν σκεφτεί κάτι αντίστοιχο. που θα έλεγα ότι στις περιοχές αυτές είναι ακόμη πιο σημαντική η μνήμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, η κυρία Γιλέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, λέει ο Μιλήτρια. Η ομάδα μας υποστηρίζει την νέα αυτή συμφωνία, την ανανέωση τέλο πάντων. Ιδιαίτερα μας βρίσκει σύμφωνους η αύξηση της τομεακής στήριξης Είναι σημαντικό να έχουμε τέτοια στήριξη και να όχι μόνο να τη διατηρούμε αλλά και να αυξάνουμε ώστε και στις περιοχές αυτές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερους πόρους, περισσότερα μέση. Είναι σημαντικό αυτό όπως είπε και η συνάδελφος ε, και στην περιοχή της χώρας των Βάσκων και σε άλλες περιοχές. Έχουμε σημαντικό στόλο 21 από τα 28 σκάφη που αναφέρονται είναι ισπανικά και επομένως ε, ως ισπανική αντιπροσωπεία έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμφωνία αυτή. Η τομεακή λοιπόν στήριξη και η ταχύτητα της εφαρμογής είναι πάρα πάρα πολύ ικανοποιητικά στοιχεία. Ο κύριος Μιανμόρ. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την ολοκλήρωση τη συμφωνία αυτή, τη ανανέωση αυτή, ε, πέραν τη τομεακή στήριξη και άλλων στοιχείων. Είναι σημαντικό αυτό το, η περιοδικότητα των 5 ετών πλέον ανανέωση και όχι 4. Δίνει μια σταθερότητα για τους τόλους, για τους αλληλείς και πρέπει να συνεχίσουμε με αυτές τις αλληλευτικές ε, συμφωνίες με τρίτες χώρες που είναι απολύτως απαραίτητες ε, για τα κράτη-μέλη αλλά και σωστή ισορροπία για τις ενεχόμενες αυτές τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γονθάλεθ και εγώ, πρόεδρε, απλώς να χαιρετήσω την ε, ολοκλήρωση συμφωνίας αυτής. Ε, πάνω από 20 σκάφη, όχι μόνο από τον Μπιλμπάο, όχι μόνο βασικά, και από τη Γαλήθεια έχουμε και από στην Ισπανία και εμείς έχουμε. Και το πρωτόκολλο αναφέρεται στα είδη που επιτρέπονται και απαγορεύεται η αλίευσή τους. Θα αποφύγουμε λοιπόν ε, επιδείνωση του αποθέματος. Ε, έχουμε μια καλή πλαισίωση. Θα έχετε τη στήριξή μας για τέτοιες συμφωνίες ελευθερικές με τρίτες χώρες που είναι εποφελής και για τις ε, δύο πλευρές. Να συμπεράνω ότι συνολικά ο Ισπανικός στόλος από όλε τις αυτόνομες περιοχές ε, θα υποφεληθεί, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, ε, τα 400, οι 400.000 πηγαίνει στην υποστήριξη του ηλεκτρικού τομέα μας, είπατε. Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι αυτοί, να σας ρωτήσω εγώ. Ε, πρόεδρε, Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, τα μέλη για τα καλά τους λόγια. Ε, προφανώς ε, πολύ σημαντικό μέρος του στόλου αυτού του ενεχόμενου είναι ισπανικός για την ε, συμμετοχή των γυναικών στον τομέα και την προώθησή του. Ε, είναι σημαντικό πράγματι και συχνά το συμπεριλαμβάνουμε. οι γυναίκες περισσότερο συμμετέχουν στη, στον μεταποιητικό τομέα, κλάδο. Αλλά δεν έχουμε εκφορτώσεις ειδικά στους άτομε και επομένως η μεταποίηση δεν ενέχεται τόσο πολύ ε, στα ποσά που δίνονται στην τομεακή στήριξη. Βεβαίω και είναι σημαντικό στοιχείο για εμάς. Ε, δεν αποκλείεται λοιπόν, εάν καθίσουμε στο τέλος του έτους, ε, στην αρχή του επόμενου έτους, να συζητήσουμε προτεραιότητες για την τομεακή στήριξη, στον τομέα της μεταποίησης παρότι εμείς δεν εκφορτώνουμε, θα σημειωθεί το θέμα των φίλων ή η συμμετοχή των γυναικών. Για την ε, μικρή σε κλίμακος αλία, σημαντικό τμήμα της στήριξης επήγαινε στην μικρή κλίμακα αλία στα προηγούμενα πρωτόκολλα, από ό,τι κατενόησα, αλλά πρέπει να σας πω ότι όταν διαπραγματευόμαστε το πρωτόκολλο δεν μπαίνουμε στα λεπτομέρειε των έργων που θα στηριχθούν, αλλά μιλούμε για ημιβιομηχανική αλληλεία από πλευρά του, αυτό μα έχουν πει, γιατί θέλουν να αναπτύξουν τι εξαγωγέ. Και επομένω η μικρή κλίμακα δεν είναι πρόβλημα. Ίσως όμως να ζητήσουν περισσότερη στήριξη για ημιβιομηχανική κλίμακα και για κάποια εργαστήρια αυτή τη στιγμή δεν μπορούν για λόγους φυτογειονομικούς να ε, εξαγάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τους ενδιαφέρει πολύ αυτό. Αυτό θα είναι επιτάπητος στις συζητήσεις του χρόνου, αλλά περιμένουμε στο παρόν γιατί χρειάζεται διάλογος για να εντοπίσει κανείς και εκείνοι τι χρειάζονται και εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Είναι αλήθεια ότι σε προηγούμενα πρωτόκολλα σημαντικό μέρος στήριξη πήγαινε στην μικρή κλίμακας αλία. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι τα μέλη για καλά τους λόγια. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Ε, το ΕΛΚ θα ορίσει εισηγητή εδώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Το απόγευμα θα έχουμε παρουσίαση για το μέλλον του αλληλευτικού τομέα, το οποίο θα θέσει τις παραμέτρους ε, για τα επόμενα πέντε χρόνια. Δεν πρέπει να το χάσετε. Τα λέμε μετά.